Καλώ Καλώς ήλθατε στο δεύτερο ημίχρονο της ε, Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων. Ξεκινάμε με την ανταλλαγή Απόψεων με την Ιλιάνα Ιβάνοβα, που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Και είναι εδώ γιατί τι θέλουμε να έρθει ενώπιόν μας και να μας παρουσιάσει σε λεπτομέρειες την ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για την εγγύηση για την νεότητα, τα πρώτα βήματα τα οποία ανελήφθησαν σε σχέση με την εφαρμογή και τους ελοχεύων κινδύνους που βρίσκονται ενώπιόν μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα και γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα που συνάπτονται με την εγγύηση για τους νέους και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και πιστεύω ότι θα μπορέσετε να μας πείτε κάτι περισσότερο για τα θέματα αυτά. Καλώς ήρθατε λοιπόν και θέλουμε να σας ακούσουμε με μεγάλη προσοχή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ <clears throat> κυρία Πρόεδρε. Είναι και για μένα μεγάλη χαρά που είμαι εδώ ενώπιόν σας. Είναι η δεύτερη φορά που παρουσιάζουμε αυτή την ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από την παρουσίαση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ για την υψή τη σημασία η Επιτροπή σα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωρίσουν την άποψή μα σε σχέση με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Το πρόβλημα τη ανεργία των νέων δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθώ και να το περιγράψω σε λεπτομέρειε. Η εγγύηση για του νέου και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων έχει σαν στόχο να δώσει σε αυτούς τους ανέργους νέους την ευκαιρία να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας και να μπορέσουν να κάνουν μια θετική συνεισφορά στην κοινωνία μας. Είναι πολυδάπανο το πρόγραμμα αυτό, αλλά δεν έχουμε και καμιά εναλλακτική λύση. Δεν θέλουμε να έχουμε το τεράστιο κοινωνικό-οικονομικό κόστος της ανεργίας, των επιδομάτων ανεργίας, των ε, φόρων που χάνονται, το κόστος αυτό υπολογίστηκε σε περίπου 153 δισεκατομμύρια το χρόνο, πάνω από 1% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της σημασίας λοιπόν του θέματος αυτού, που επηρεάζει τα περισσότερα κρατημένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν απαραίτητο για μας να μπορέσουμε σε πρώιμο στάδιο να παρέμβουμε και να δώσουμε στους λήπτες αποφάσεων μια <clears throat> σαφή και έγκαιρη άποψη σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό για την εγγύηση για τους νέους. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να επιτύχει το πρόγραμμα αυτό, αλλά ως ελεκτικός φορέας. Θέλουμε να σας δώσουμε μια αντικειμενική ε, εικόνα σε σχέση με το πώς βλέπουμε για αυτό το, αυτό το πρόγραμμα και πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Εγώ συμμερίζω με τις περισσότερες απόψεις που ακούστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια σε μια συζήτηση με το Συμβούλιο. Πιστεύω ότι το, η πρωτοβουλία για τους νέους και η εγγύηση για τους νέους δεν είναι πανάκια μένα, αλλά είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να συνοδεύεται από οικονομικά μέτρα τα οποία υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Το σύστημα εγγύησης δίνει μια βραχυπρόθεσμη υποστήριξη για τους νέους, αλλά μας ενδιαφέρει να μπορούμε να έχουμε τις μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές αλλαγές στα κάτι μέλη για να εξασφαλίσουμε καλύτερη μετάβαση από το σχολικό σύστημα στο χώρο εργασίας και να αποφύγουμε ότι οι νέοι μένουν στο περιθώριο. Η έκθεσή μα αξιολόγησε το κατά πόσο οι υπηρεσίε τη Κομισιόν έχουν δώσει την απαραίτητη υποστήριξη στα κρατη για να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτό το σύστημα υγεία για του νέου και εντοπίσουν του δυνητικού κινδύνου οι οποίοι συνάπτονται με την εφαρμογή του προγράμματο αυτού. Αυτό το οποίο εμεί διαπιστώσαμε είναι ότι γενικά η Κομισιόν έχει δώσει επαρκή και έγκαιρη βοήθεια στα κρατη για να εφαρμόσουν αυτά τα προγράμματα, μέσα βέβαια στα προγράμματα που έχει θέσει η σύσταση του Συμβουλίου, παραδείγματο χάρη η Κομισιόν έδωσε κατευθυντήρες γραμμές στα κάτι μέλη για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων αυτών πέντε μήνες, μέσα στους πέντε μήνες που ακολούθησαν την σύσταση του Συμβουλίου και έκανε πλήρες και έγκαιρες ε, ε, επισκοπήσεις του τρόπου εφαρμογής και εντόπισε πολλά από τα σημεία <clears throat> όπου παρουσιάστηκαν ελλείψεις και προβλήματα. Τρεις πτυχέ όμως δεν τις αντιμετώπισε η Κομισιόν σε σχέση με την ε, πληροφορική και τις ψηφιακές ε, δεξιότητες και τη δυνατότητα ε, αλληλομάθησης κατά κάποιο τρόπο μεταξύ των νέων. Τα κρατημένη επίσης έχουν μεταρρυθμίσει σε κάποιο βαθμό τις ε, προτάσεις τους μετά από αυτά που είπε η Κομισιόν. Έχουμε εντοπίσει τρεις κύριους κινδύνους σε σχέση με το επαρκές της χρηματοδότηση σε σχέση με την καλή ποιότητα των προσφορών προς τους νέους και τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν εποπτεύει και αναφέρει για τα αποτελέσματα αυτού του σχεδίου. Για το επαρκές χρηματοδότηση πρώτα απ' όλα. Ακόμα και η κλίμακα του προγράμματος θεωρούμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά ο σχεδιασμός και η κλίμακα του προγράμματος αυτού. Μέσα στο πρόγραμμα 2014 ως 2020 θα έχει χρηματοδότηση 24,7 δισεκατομμύρια από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Κοινωνικό Ταμείο η πρωτοβουλία αυτή, αλλά θα χρειαστούν πρόσθετα κονδύλια για τα πιο βραχυπρόθεσμα μέτρα για τους άνεργους νέους και για να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι διαφορετικές αλλαγές σε τομείς όπως είναι η κατάρτιση, η αναζήτηση εργασίας και τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών. Είδαμε ότι δεν υπήρχε κάποια ε, αξιόπιστη εκτίμηση του κόστους για το σχέδιο αυτό, για την εγγύηση για τους νέους. Κανένα από τα κράτη που μας έδωσαν στοιχεία δεν μας έδωσε στοιχεία για το κόστος εφαρμογής των διαθωτικών αλλαγών που απαιτούνται. Βάσει της άποψης της Κομισιόν, εννέα κράτη-μέλη δεν έχουν δώσει καθόλου στοιχεία σε σχέση με τα εθνικά προγράμματα και την ανάγκη χρηματοδότησης. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για μας είναι το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν έχει εκτελέσει τις απαραίτητες εκθέσεις αντικτύπου προτού εφαρμόσει αυτή την εγγύηση. Έχουμε μονάχα τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Οπότε ξέρουμε ότι τα μόνα αριθμητικά στοιχεία τα οποία υπολογίζουν το κόστος το ετήσιο του προγράμματος αυτού, ενός προγράμματος το οποίο θα ήταν λειτουργικό σε περίπου 21 δισεκατομμύρια ευρώ το, χρώμα, το χρόνο, ενώ εμείς έχουμε 24,7 για μια ετία. Εν κατακλείδη είδαμε ότι υπάρχουν ανεπαρκείς πληροφορίες διαθέσιμες σε σχέση με το συνολικό κόστος του προγράμματος αυτού και αυτό μπορεί να υποσκάψει την σωστή εφαρμογή και το τελικό αντίκτυπο του προγράμματος που αφορούν εκατομμύρια ανέργων στην Ευρώπη. Ο δεύτερος κίνδυνος έχει να κάνει με τον με την έλλειψη προσδιορισμού του τι σημαίνει μια προσφορά υψηλής ποιότητας. Αυτό βρίσκεται στην ε, καρδιά του προγράμματος. Η πρόβλεψη είναι ότι όλοι οι νέοι μέχρι 25 ετών θα πρέπει να έχουν μια καλή προσφορά, καλής ποιότητας προσφορά μέσα σε τέσσερις μήνες από τη στιγμή που φεύγουν από το εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά δεν υπάρχει καμία σαφής διευκρίνηση του τι είναι μια προσφορά υψηλή ποιότητα, καλή ποιότητα και ούτε αναφέρεται ποιο είναι υπεύθυνο για να το εξασφαλίσει αυτό. Θεωρούμε ότι η ποιότητα τη προσφορά που είναι προ του νέου είναι ένα κύριο στοιχείο χωρί μια σειρά από χαρακτηριστικά όπω είναι το είδο συμβολέου, διάρκεια, ε, αποδοχές σε σχέση με το κόστο, διαβίωση κτλ. Υπάρχει κίνδυνο τα τη μέλη να δώσουν στους νέους ε, θέσεις που δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τι μεσοπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές εργασίες. Εν καιρό αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη αποτελεσματική εφαρμογή και όχι συνεκτική ε, εφαρμογή μεταξύ κρατών μελών. Το τρίτο και όχι το υποδέστερο στοιχείο κινδύνου είναι το σύστημα απόδοσης αναφορών και εκθέσεων το οποίο είναι ακόμα υπό προετοιμασία. Για να έχουμε μια σαφή εικόνα της ε, εφαρμογής του συστήματος αυτού και του σχεδίου θέλουμε να υπάρχει σωστή διαχείριση ώστε να μπορούμε να δρούμε προδραστικά και να βοηθούμε τους νέους. Εμείς διαπιστώσαμε ότι οι ρυθμίσεις για πλήρη παροχή εκθέσεων δεν είχαν ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του προγράμματος αυτού από την αρχή. Υπάρχουν κάποιες ε, ρήτρε σε σχέση με το ε, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, την Επιτροπή Απασχόλησης του Συμβουλίου, αλλά τη στιγμή που κάναμε τον έλεγχο ως ελεγκτικό συνέδριο, βρήκαμε ότι δεν υπήρχαν σχέδια να υπάρχουν εκθέσεις για, τα, για την πρόοδο του σχεδίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά από την δημοσίευση της έκθεσής μας όμως σημειώνουμε ότι η Κομισιόν αποφάσισε να έρχεται ενώπιον του Κοινοβουλίου και να σας δίνει εκθέσεις για την πρόοδο που επιτελείται. Εν κατακλείδη θα ήθελα να πω και κάτι για τις δικές μας συστάσεις. Επί τη βάση των πορισμάτων μας κάνουμε τρεις ε, συστάσεις που κατά την απόψή μας θα βοηθήσουν ιδιαίτερα την σωστή εφαρμογή της εγγύησης για τους νέους. Η πρώτη αφορά τη χρηματοδότηση. Εμείς συνιστούμε τα κράτη-μέλη να δώσουν μια πλήρη απεικόνηση του κόστους όλων των μέτρων που αφορούν την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, ώστε η Κομισιόν μπορεί να αξιολογήσει το επίπεδο της απαιτούμενης χρηματοδότησης η δεύτερη μας σύσταση είναι να βελτιωθεί η φύση των προσφορών προς τους νέους σε ό,τι αφορά την ποιότητά τους. Θέλουμε η Κομισιόν να παρουσιάσει μια σειρά από χαρακτηριστικά που συγκροτούν την ποιότητα των προτινομένων θέσεων εργασίας και μαθητιών και αυτό θα μπορούσε να βασίζεται σε στοιχεία που να καθορίζουν τι είναι η καλής ποιότητος ε, εργασία μέσα στι κατευθυντήρε γραμμέ τη Κομισιόν. Και το τρίτο σημείο έχει να κάνει με την παροχή εκθέσεων. Εμεί θέλουμε και πάλι να συζητήσουμε στην Κομισιόν να δημιουργήσει ένα πλήρε εποπτικό σύστημα για την ε, πρωτοβουλία για του νέου που να καλύπτει και τι απαραίτητε διαθωτικέ αλλαγέ και τα μέτρα τα οποία στοχεύουν συγκεκριμένα άτομα. Και επίση ζητούμε όλα αυτά να την χάνουν αναφορών όχι μόνο προ το Συμβούλιο αλλά και προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπω είπα προηγουμένω τρέφουμε τις ελπίδες ότι θα είναι επιτυχής η εγγύηση για και όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τα κρατη θα πρέπει να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους και να μπορέσει να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα του το να δυνατό. Χρησιμοποιώ επίσης αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την επικοδομητική τη στάση και τη συνεργασία που έδειξε προς τα άλλα θεσμικά όργανα και θέλω φυσικά να ευχαριστήσω και εσάς την Επιτροπή σας και εσάς κυρία Πρόεδρε που με, καλέσατε, με προσκαλέσατε εδώ και προσβλέπω στα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την ε, ε, εισαγωγή. Μπορείτε τώρα να κάνετε ερωτήσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε με τους, με τους εισηγητές για το θέμα της πρωτοβουλίας των νέων. Πρώτα η κυρία Μωρέν Σαρτή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ ε, την κυρία Ιβάνοβα που ήρθε να μας κάνει μια παρουσίαση για αυτήν την έκθεση την πολύ σημαντική είναι η δική σας ε, θεώρηση των πραγμάτων για την εγγύηση για την νεολαία και την ε, πρωτοβουλία για τους νέους. Εγώ διάβασα την έκθεσή σας, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ήταν, όμως έχω κάποιες παρατηρήσεις το έχουμε συζητήσει άλλωστε και άλλες φορές οι δυο μας για το πώς μπορούμε να εμβαθύνουμε ε, και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το μηχανισμό. Το πρώτο πράγμα που διαπιστώνει κανείς επιτόπου είναι η τεράστια σύγχυση που υπάρχει στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ κρατών, των κρατών μελών ε, μεταξύ της εγγύησης για την νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων είναι κάτι το πολύ επιβλαβές αυτό, γιατί τελικά η προσπάθεια επικοινωνία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων κατά κάποιο τρόπο ε, καπέλωσε το στόχο ε, που θέλαμε να έχουμε ότι δηλαδή αυτή η πρωτοβουλία θα έπρεπε να στοχεύει κυρίως στους, στην ανεργία των νέων. Δηλαδή αυτό που θέλαμε είναι στόχευση περισσότερο των ε, περιοχών όπου ε, άτομα 15 με 25 ετών ε, εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά ανεργίας και έχει υπάρξει μία σύγχυση μεταξύ αυτών των δύο και νομίζω ότι για το πρώτο από τα δύο που ανέφερα είναι το, το θέμα της επικοινωνίας. Εκεί πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ αυτή την πολιτική της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Είδατε, τα μπερδεύω κι εγώ τελικά. Ας τα ξαναπώ. Λοιπόν, πρώτον έχουμε το θέμα της εγγύησης για την νεολαία και μετά την ενίσχυση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Είναι πολύ επιβλαβής αυτή η σύγχυση γιατί τουλάχιστον στα μέρη όπου πηγαίνω εγώ, όχι μόνο στη χώρα μου αλλά και σε άλλες χώρες, όπου πηγαίνω διαπιστώνω ότι ε, οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων δεν καταλαβαίνουν ακριβώς πώς τοποθετούνται μεταξύ αυτών των πολιτικών. Και η επικοινωνία για την πρωτοβουλία, για την απασχόληση των νέων, αμβλύνει κάπως ε, την πολιτική μας για τις εγγυήσεις για την νεολαία. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα ε, να ε, σας ζητήσω να σχολιάσετε εκτός από τη σύγχυση είναι η αναγκαιότητα ύπαρξης ε, προγραμμάτων. Το καταλαβαίνω και συμμερίζομαι τη βούλησή σας να να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει μια καλή αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που διατίθενται, αλλά δεν υπάρχουν προγράμματα αυτή τη στιγμή σήμερα. Είναι πολλά τα χρόνια από τότε που κάναμε τη διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για ε, την εγγύηση για, τις, ε, την νεολαία και δεν υπάρχουν προγράμματα να την υποστηρίξουν. Αυτό είναι το δεύτερο που θα ήθελα να πω λοιπόν, πώς μπορούμε να, να προωθήσουμε τέτοιου είδους προγράμματα. Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να θέσω είναι το εξής αγωνιστήκαμε πάρα πολύ ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ε, να υπάρξει 20% που θα διατίθεται για την καταπολέμηση της ένδυας. Ε, επομένως, η ένδυα μεταξύ των νέων η άποψή σας, η ανάλυση, της, ε, η ανάλυση οικονομική που κάνετε και μας μας ενδιαφέρει επίσης πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε να ε, μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε αυτά τα προγράμματα τα οποία ιδιαίτερα στοχεύουν την καταπολέμηση της ένδυας των νέων. Και τέλος, δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω πολύ περισσότερο, αλλά πραγματικά εγώ προσδοκώ πάρα πολλά από τη συζήτηση αυτή. Είπατε ότι αυτή η πολιτική αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Εγώ δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι αν πάει κανείς επιτόπου να δει τι γίνεται, είναι σε εμβριακό στάδιο. Έχουμε πολύ διαφορετικές ταχύτητες ακολουθήσει ε, σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών. Θελήσαμε πραγματικά να επιταχύνουμε με το Συμβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, την οποία χαιρετίζω βεβαίως ε, σήμερα. Αλλά πραγματικά πρέπει να ακολουθήσει και να ακολουθήσει και το τοπικό επίπεδο όλα αυτά τα πράγματα, που είναι κάτι που δεν γίνεται. Συμφωνώ λοιπόν απολύτω με αυτό που είπατε για, για την καλή τη ποιότητα προσφορά ε, στην εκπαίδευση, στη μαθητεία, ε, στην ε, άσκηση. Καταλαβαίνω ότι αυτό που είπατε για τον ορισμό της καλής ποιότητας προσφοράς, δεν είναι ίδιος ο ορισμός για όλα τα επίπεδα. Έχουμε νέους που βγαίνουν, ε, που δεν έχουν δεξιότητες, που δεν έχουν επαγγελματικά προσόντα. Έχουμε νέους που έχουν ε, κάποιο δίπλωμα. Ε, δεν είναι το ίδιο δεν είναι ε, οι ίδιες οι, οι προσδοκίες κάθε φορά ανάλογα με τους νέους για τους οποίους μιλάμε. Και συνεπώς είναι διαφορετική και η αντίδρασή μας προκειμένου να τους βοηθήσουμε. Δεδομένες λοιπόν της ποικιλομορφίας που εμφανίζουν αυτοί οι νέοι πληθυσμοί που μπορούν να επωφεληθούν από αυτή την πολιτική, πρέπει να μην, είμαστε, να μην έχουμε στέγανα, πρέπει να μπορέσουμε να επαγρυπνούμε ώστε να εξασφαλίζουμε ότι αυτές οι πολιτικές που είναι μακροχρόνιες, βαριές ε, ε, πολιτικές και με δύσκολο κοινό, Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τις φέρουμε εις πέρας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ε, σας ε, ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τώρα με τους ε, σκιώδεις ε, εισηγητές, καταρχήν από την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ το ελεγκτικό συνέδριο, την κυρία Ιβάνοβα για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης. Ε, το χρειαζόμασταν οπωσδήποτε από τη στιγμή που είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε αυτό το πρόγραμμα από τότε που ετέθησε σε ισχύ. Είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων. Θέλαμε να γνωρίζουμε τι λειτουργεί και τι όχι. Ε, ένα ανεξάρτητο σώμα, το ελεγκτικό συνέδριο, εμπλουτίζει τη συζήτηση και μας βοηθάει στο να μην είμαστε πολιτικά τουλάχιστον προκατηλημένοι. Πρέπει να υπάρχει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση που να αφορά την εγγύηση για τους νέους και νομίζω ότι το έγγραφο που μας έχει κατατεθεί εξυπηρετεί αυτό το στόχο. Οι τρεις συστάσεις ε, που στάλησαν στην Επιτροπή αυτές τις ε, συμμεριζόμαστε πράγματι πρέπει να υπάρχει σαφήνεια από τα κράτη-μέλη κυρίως όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πάνω απ' όλα είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει εγγυημένη ποιότητα των ε, προτάσεων. Ε, στην εγγύηση αυτή δεν μπορούν να υπάρχουν ε, καταχρήσεις, δεν θα πρέπει αυτά τα στάζ και η μαθητεία να είναι ο προθάλαμος των επισφαλών θέσεων εργασίας. Νομίζω ότι είναι ακόμα λιγάκι νωρίς για να τριαμβολογούμε. Αυτό αυτό που μπορεί να βελτιωθεί, θα έλεγα με ικανοποιητικό τρόπο, είναι το ε, ποσοστό απασχόλησης των νέων. Η δική μου χώρα, η Ιταλία, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Δυστυχώς η ε, ανεργία των νέων εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή και αυτό δείχνει κάτι ε, που είναι σαφές σε σχέση με την εγγύηση των νέων. Αυτό δεν είναι ένα εργαλείο απλά και μόνο για να υπάρχουν θέσει απασχόλησης. Ε, σαφώς και να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη ή καταπολέμηση ενεργείας, αλλά να υπάρχουν επενδύσεις σε στρατηγικούς ε, τομείς όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, οι ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και όλα τα άλλα. Επίσης, να υπάρχει μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το πλήρες δυναμικό. Όπως σας είπα υπάρχουν διάφορα προβλήματα, ε, πολύ περίπλοκα στα κράτη-μέλη ε, και έτσι από την υπερβολική γραφειοκρατία μπορούμε να περάσουμε την ε, λεπτομερή καταγραφή των ε, προγραμμάτων, ούτε και αυτό είναι θετικό. Και προστίθεται το ότι πάρα πολλοί νέοι, κυρίως αυτοί που το χρειάζονται, δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη της εγγύησης ε, των νέων και την πρωτοβουλία για την ανική απασχόληση. Άρα είναι απαραίτητο για όλους τους δημόσιους θεσμούς να γίνει γνωστή αυτή η πρωτοβουλία και αυτό θα εξυπηρετήσει πάνω απ' όλα στο να δείξουν τα κράτη-μέλη την πολιτική βούληση να επενδύσουν στους νέους και επίσης ε, να κάνουν τα πάντα για τη γενιά μας, ξεκινώντας από την χρηματοδότηση αυτής της εγγύησης ε, μέχρι και την πρωτοβουλία κατά τα επόμενα έτη, ε, να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων σε συνδυασμό με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί πρέπει, και ένα πράγμα πρέπει να διασφαλίσουμε, ότι θα είναι πράγματι εγγυημένη η εγγύηση για τους νέους από τους συντηρητικούς και τους ε, μεταρρυθμιστές. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Η κυρία Ζητνάσκα. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ιβάνοβα για αυτή την έκθεση, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμη και όπως αναφέρθηκε ήδη, δεν είναι όλα απόλυτα σαφή και δυστυχώς ε, ε, δεν τα γνωρίζουν τόσο καλά και τα κράτη Εγώ ε, προέρχομαι από τη Σλοβακία και θέλω να σας πω ότι στη Σλοβακία υπάρχει ένα μεγάλο κενό κυρίως όσον αφορά τη χρήση των κοντιλίων και τον έλεγχο όσον αφορά την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων. Ε, επ' αυτού θα ήθελα να συνεχίσω να εργάζομαι, συνεργάζομαι με το Υπουργείο μας ε, για θέματα εργασίας και απασχόλησης, έτσι ώστε τα κονδύλια που εκταμιεύονται να χρησιμοποιούνται σωστά στην Σλοβακία γιατί νομίζω ότι αυτή είναι μια τελευταία ευκαιρία για να σώσουμε μια ολόκληρη γενιά νέων και γνωρίζουμε ότι όταν οι νέοι μετά το πανεπιστήμιο δεν βρίσκουν εργασία αυτό σημαίνει ότι ε, θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον ε, πολλά προβλήματα και αυτό θα είναι εις βάρος του συνόλου της ε, κοινωνίας. Όπως λοιπόν ήδη αναφέρθηκε στις συστάσεις που κάνατε, είπατε πολλά θετικά στοιχεία, εμείς τα προσυπογράφουμε και θέλω να σας πω ότι πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα της ε, προσφοράς. Αυτό που είπε η κυρία Μωρόν Σαντιέ και συμφωνώ απόλυτα. Ίσως ε, να μην ενδείκνεται πλήρως να υπάρχει ε, ένας ενιαίος ορισμός της ποιοτική απασχόλησης. Εσείς μιλήσατε ήδη ε, για, το, για ποια κριτήρια πρέπει να συζητάμε. Να συζητήσουμε με λεπτομέρειες για την κατάσταση των νέων ποικίλη και έτσι λοιπόν η κατάσταση ε, θα πρέπει να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Τα μέτρα αναδιάρθρωσης μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα. Και ίσως μπορείτε να μας πείτε περισσότερα να μας εξηγήσετε την άποψή σας ε, το τι μορφή θα λάβει αυτή η ποιοτική προσφορά. Επίσης θα ήθελα να έχω ένα, να υπογραμμίσω έναν καλύτερο έλεγχο και ε, το πώς ε, θα χρησιμοποιούνται αυτά τα κονδύλια. Γιατί εμείς είμαστε μάρτυρες και αυτού και άλλων προγραμμάτων όπου ε, τα οικονομικά μέσα δεν ε, χρησιμοποιούνται όπως πρέπει. Θα ήταν λοιπόν κρίμα αν και σε αυτό το πρόγραμμα δεν επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Ελπίζω λοιπόν και η δική μας η Επιτροπή να συμβάλλει έτσι ώστε να ε, διαφυλάξουμε καλύτερα τα κονδύλια του Ευρωπαίου Φορολογούμενου. Ε, μήπως εκπροσωπείτε εσείς τους φιλελεύθερους. Μάλιστα, εγώ είμαι από τους ε, φιλελεύθερους. Δεν έχω συμφωνήσει με τη Μαρτίνα να μιλήσω εκ μέρους της, αλλά θα ήθελα να φέρω τρία μικρά σημεία. Πρώτον, η μελέτη αντικτύπου. Για να γίνει αυτή χρειαζόμαστε κάποια ε, κριτήρια και η ανεργία των νέων είναι ένα εξ αυτών. Επίσης ε, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία στην έκθεση κομισιών, αλλά τα στατιστικά δεδομένα από μόνα τους ε, δεν λένε την αλήθεια. Πρέπει να αναλυθεί το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο. Στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη, ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της χρήσης των κονδυλίων. Εγώ είμαι από την Εστονία, εμείς δεν έχουμε τόσο υψηλό ε, ποσοστό ανεργία στους νέους για ένα και πλέον μόνο λόγο γιατί έχουν φύγει από τη χώρα, δεν είναι εκεί, δεν υπάρχουν. Κάτι άλλο. Ε, η ανεργία και η πρωτοβουλία σε εμά είναι όπως σας είπα χαμηλότεροι. Οι μεγάλες χώρες ε, κατά κανόνα έχουν μια διαφοροποιημένη προσέγγιση. Δυστυχώς πολλές περιφέρειες δεν ε, ε, υποφελούνται. Και υπάρχει αυτός ο φόβος και για τις μικρότερες χώρες. Στην Εστονία, παραδείγματο χάρη, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποιημένη προσέγγιση ανάλογα με την περιοχή. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές όπου η ανεργία των νέων είναι 25% αλλά και μεγαλύτερη ίσως, όχι όμως η ανεργία δεν είναι τόσο ψηλή στο σύνολο της χώρας, είναι χαμηλότερη και αυτό είναι κάτι που ίσως θα πρέπει να το σκεφτούμε. Από την ΚΟΕ παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση από το ελεκτικό συνέδριο. Αν είχαμε λάβει υπόψη μας όλα αυτά τα στοιχεία, θα ήταν αρκετά διαφορετικό το πρόγραμμα από αυτό που είναι τώρα και θα είχε διαφορετικά μέτρα από αυτά τα οποία προβλέπονται αυτά στιγμή μέσα στο πρόγραμμα και από το Κοινωνικό Ταμείο. Εγώ ως Πορτογαλέζα Βλέπω ότι υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία στην Πορτογαλία σε σχέση με την εκτέλεση αυτού του σχεδίου και σε σχέση με τις ε, μορφές απασχόλησης οι οποίες θα καλυφθούν από το πρόγραμμα αυτό. Και δεν ξέρω αν υπάρχει πραγματικά κάποια ουσιαστική διαφορά σε σχέση με αυτά τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι, ότι μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπήρξαν πολλά στάσμα μαθητείας, πολλά προγράμματα εισαγωγής επιχειρήσεις και το θέμα είναι από έποψη ποιότητας τι καινούριο μας φέρνει αυτό το πρόγραμμα. Φέρνει κάτι ή δεν φέρνει κάτι. Έχουμε ένα γιγάντιο πρόβλημα η Κομισιόν κανονικά πρέπει να αναλάβει την ευθύνη αυτού του προγράμματος, αλλά φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε αναλάβει ως κάτι μέλη μια σειρά από πειράματα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και ουσιαστικά καλύπτονται τα προβλεπόμενα αυτά κονδύλια και τις απασχόλησης από πιο φτηνά προγράμματα και δεν έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα τα προγράμματα αυτά παρά μόνο να αυξάνουν το συνολικό κόστος. Μιλάμε για δημιουργία μόνιμων θέσεων απασχόλησης αλλά δεν εξασφαλίζουμε την κάλυψη αυτών των θέσεων απασχόλησης. Όταν εσείς λοιπόν κάνετε συστάσεις και πολύ καλό είναι αυτό που κάνετε για τα κριτήρια ποιότητας σε επίπεδο απασχόλησης πέραν της διάρκειας του συμβολέου που λαμβάνει ένας νέος, πέραν της ποιότητας της κατάρτισης, είναι σημαντική η ίδια η θέση ούτε καν και η αμοιβή είναι τόσο σημαντική. Για μένα αυτό που προέχει είναι η ποιότητα της θέσης απασχόλησης, ότι αυτά τα άτομα έχουν την εξασφάλιση όλων των κοινωνικών δικαιωμάτων τους, με τον ίδιο τρόπο που έχει οποιοδήποτε άλλος απασχολούμενος. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε άλλου είδους εργασίας, διαφοροποιημένη μορφή εργασίας με, λιγότερες, με λιγότερα κοινωνικά δικαιώματα βάσει νέων ειδών συμβολέων. Θα πρέπει λοιπόν, α, γι' αυτό κάναμε ορισμένε προτάσει τροπολογία στον κανονισμό που δυστυχώ το Κοινοβούλιο δεν δέχτηκε. Και σε σχέση με την αμοιβή των νέων, η αμοιβή αυτή θα πρέπει να βρίσκεται με το, στο ίδιο επίπεδο με την αμοιβή των εργαζομένων στον αντίστοιχο τομέα. Και ανησυχώ πάρα πολύ για την απάντηση μας δίνει η Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Νομίζω θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κριτήριο ποιότητος για την ε, απασχόληση και θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά θα εξαρτηθούν πολύ από το γενικό πλαίσιο στο οποίο θα τεθεί αυτή η εργασία ποιότητος. Για να είναι εργασία ποιότητος θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του τωρινού οικονομικού κλίματος το οποίο έχει σαν στόχο να μειώσει το επίπεδο ποιότητος της εργασίας και δικαιωμάτων των εργαζομένων. Πρέπει λοιπόν μέσα σε αυτό το οικονομικό πλαίσιο να έχουμε μέτρα τα οποία θα είναι υπέρ των εργαζομένων. Δεν πρέπει λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε ως ένα πρόσχημα αυτό για να υποβαθμίσουμε ακόμα περισσότερα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το κοινοβουλίο μας λοιπόν θα πρέπει να πιέσει την Κομισιόν ώστε να προβεί το ταχύτερο δυνατό στον καθορισμό των δικτών για μία εργασία ποιότητος και να εκμεταλλευτεί και την ε, αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για να δώσει επιτέλους στο πρόγραμμα αυτό τα απαραίτητα κονδύλια ώστε για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις εκτιμήσεις που έχει κάνει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας σε σχέση με τα ποσά τα οποία απαιτούνται. Δεν ξέρω λοιπόν τι πιστεύετε κι εσείς ότι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά θα πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα για να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι συστάσεις να μην παραμείνουν άσκηση επιχάρτου και να έχουν κάποια αποτελέσματα σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό, ώστε το πρόγραμμα αυτό να είναι άξιο του ονόματός του. Λάουρα from EFTD. κυρία Άγγια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου για το έργο που έχει φέρει σε πέρας, γιατί για πρώτη φορά βλέπουμε ότι <clears throat> υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τα προβλήματα και δεν είναι απλώς εξωγήινε. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι καταλαβαίνουν τα προβλήματα, ιδίως τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εμείς στην Ιταλία. Αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων στη δική μου χώρα, το αποτέλεσμα είναι μηδενικό. Έχουν αποτύχει τα πάντα. Η εγγύηση για τους νέους, η εγγύηση για την απασχόληση των νέων. Η μεγάλη αυτή η ευκαιρία η οποία παρουσιάστηκε ως πανάκια για να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας, όπως το ανέφερε ένας πρώην Ιταλός Πρωθυπουργός, που είπε θα δημιουργηθούν δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας, μετά από δύο χρόνια ούτε 20.000 θέσεις εργασίας δεν έχουν δημιουργηθεί χάρη στο πρόγραμμα αυτό εγγύησης των νέων. Λοιπόν, μιλάμε για μια πλήρη αποτυχία. Αυτά που διαβάζω στον Ιταλικό τύπο είναι ότι οι νέοι οι οποίοι είναι στην Ιταλία είναι 52%. Αυτό είναι ντροπή, είναι όνειδος για όλους. Και το μεγαλύτερο σφάλμα, πέραν της αδυναμίας σωστής χρήσης των πόρων, γιατί αυτό είναι για μένα κάτι το δεδομένο το ότι η κυβέρνησή μου δεν μπόρεσε να υλοποιήσει προγράμματα τα οποία είναι αποτελεσματικά πέραν όμως αυτής της αποτυχίας αν συνεχίσουμε να διαπράττουμε τέτοιου είδου σοβαρά σφάλματα αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχει καμία μορφή εποπτείας. Υπάρχει απόλυτα αναποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των νέων. Κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι οι νέοι που χρειάζονται βοήθεια, τι είναι τα προγράμματα αυτά, τι είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να οργανωθούν, πώς θα πρέπει να οργανωθεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση των νέων. Δεν υπάρχει καμία παρακολούθηση για το πώς κατανέμονται τα ποσά των κονδυλίων, πώς κατανέμονται μεταξύ των διαφόρων περιοχών. Δεν είναι καμιά προσπάθεια να καταλάβουμε τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και να κάνουμε σχέδια τα οποία μπορούν να ε, κινητοποιήσουν το δυναμικό των νέων. Εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τη δράση μας είναι μια αλαζονική επιφανειακότητα. Θα πρέπει να έχουμε την ευφυΐα και την ικανότητα να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιο προϊόν το οποίο μπορούμε να το δώσουμε στους νέους. Το να έχουμε σε μια πόλη 50.000 ε, πολιτών 20 θέσεις εργασίας που προσφέρουμε στους νέους, αυτό είναι ντροπή. Στην Ιταλία λοιπόν αυτή ήταν η πραγματικότητα της εγγύησης για των νέων. Γι' αυτό εγώ περιμένω η προχρηματοδότηση η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ως σύνθημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα πρόσθετα αυτά 2 ε, δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να δαπανηθούν με ένα σωστό τρόπο. Αλλά για μένα έχει μεγάλη σημασία να ξέρω η δική μου κυβέρνηση πώς δαπάνησε μέχρι την τελευταία δεκάρα τα χρήματα που είχε πάρει για το πρόγραμμα αυτό, γιατί ξέρω ότι οι νέοι στη χώρα μου εξακολουθούν να είναι άνεργοι, να ζουν με τους γονείς τους χωρίς καμία, ε, χωρίς καμία θέση εργασίας και ουσιαστικά έχουν σπαταληθεί όλα αυτά που σας ευχαριστώ. Δύο ακόμη συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Μπορούμε να τους ακούσουμε και μετά να απαντήσετε σε όλους μαζί. Ωραία, η κυρία Μάκιντάιρ. Και μετά ο κύριος ε, Λόπες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ομάδα μας πάντα πίστευε στη δημοσιονομική πειθαρχία και στην, στον καθορισμό των πολιτικών βάσει αποτελεσμάτων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η έκθεση. Είναι σημαντικό τμήμα της δουλειάς μας ε, στην Επιτροπή μας. Είναι σημαντικό να γίνεται μία ε, επισκόπηση του πώς έχουν δαπανηθεί τα χρήματα και τι έχει επιτευχθεί γιατί αν ε, τα αποτελέσματα που είχαμε ε, σχεδιάσει δεν ε, έχουν επιτευχθεί, πρέπει να βρούμε καλύτερους τρόπους, άλλους τρόπους να επιτύχουμε τους στόχους μας. Οπότε, είμαι ευγνώμων στην κυρία Ιβάνοβα που είναι εδώ σήμερα και που παρουσίασε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Πολλές ανησυχίες έχω σε σχέση με αυτά που μας είπατε ως πορίσματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου και δεν είπε ποιο είναι το αναμενόμενο κόστος και από το αποτέλεσμα. Γιατί αυτό, ε, και αυτό είναι τμήμα της διαδικασίας για, τις, ε, για όλες τις μεγάλες ε, πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε αυτό είναι ήδη προβληματικό. Αν θέλουμε να παρακολουθούμε σωστά, πρέπει από την αρχή να ξέρουμε τι θέλουμε να επιτύχουμε. Στην πρώτη σας σύσταση λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να παρέχουν σαφή και πλήρη επισκόπηση του κόστους όλων των προγραμματισμένων μέτρων για την καταπολέμηση της ενεργείας κλπ. κλπ. Δεν είναι μόνο το κόστος. Πρέπει να μπορούμε να καταλάβουμε και τα ωφέλη και από ποσοτική και από ποιοτική απόψεως. Αν δεν πούμε τι θέλουμε να επιτύχουμε, πώς μπορούμε να ε, να δούμε μετά κατά πόσο ε, τα επιτύχαμε ή όχι. Και στο τέλος της τρίτης σας ε, σύστασης είπατε ότι τα αποτελέσματα της παρακολούθησης πρέπει να υποβάλλονται στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Κάποιος θα έλεγε ότι αυτό είναι αυτονόητο. Όχι βέβαια, δεν συμβαίνει αυτό και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που λέει στην παράγραφο 68 στις παρατηρήσεις σας που αναφέρεται ότι δεν υπάρχει τέτοιο, ε, δεν έχει προγραμματιστεί τέτοιου είδους ε, υποβολή εκθέσεων στο Κοινοβούλιο και νομίζω ότι ως Κοινοβούλιο θα έπρεπε να ζητούμε η παρακολούθηση αυτή της εφαρμογής και η εποπτεία των επιτευγμάτων να αποτελεί αντικείμενο έκθεση που θα υποβάλλεται σε μας. Γιατί εμείς πώς ως εκπρόσωποι όλων αυτών των νέων που είναι άνεργοι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι επιτυγχάνουμε και τι όχι. Παρά το ότι έχουμε αυτή την πρωτοβουλία για την νεολαία, για την απασχόληση των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη, πρέπει να συνεργαστούμε ε, και να προσαρμόζουμε με τα διάφορα κράτη-μέλη τις λύσεις, γιατί δεν θα βρούμε ποτέ μια λύση που να ταιριάζει σε όλα τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι καλύτερα βρίσκει κανείς και εφαρμόζει πολιτικές σε επίπεδο κράτους-μέλους ε, και το λέω αυτό και από απόψε ως ε, και από απόψε ε, αποτελεσμάτων. Όσον αφορά λοιπόν την παρακολούθηση και την ειδική ανάλυση που μπορεί να γίνει, νομίζω ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε καλύτερα τις ε, βέλτιστες πρακτικές μας και να καταλάβουν και τα κράτη-μέλη τι επιτυγχάνουν και τι όχι. Πάρα πολύ χαίρομαι που άρχισαν 2,2 εκατομμύρια μαθητείες στο Ηνωμένο Βασίλειο το περασμένο έτος, αλλά τι να σας πω, δεν μπορώ να πω ότι εφησυχάζω, γιατί εγώ βλέπω ότι στην εκλογική μου περιφέρεια αυξάνεται ακόμη η ανεργία. Δεν είναι λοιπόν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να, πει, να κάνει μάθημα στην υπόλοιπη ε, Ευρώπη. Πρέπει νομίζω να δούμε πώς, τι δουλεύει και πώς μπορούμε να το ε, αξιοποιήσουμε αυτό που λειτουργεί καλύτερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε δηλαδή τι περιπτώσει όπου η καλή επένδυση είχε, έχει επιφέρει καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Πάρα πολύ χρήσιμη ήταν αυτή η εκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Λόπελ από την ομάδα των σοσιαλιστών. Και μετά μπορείτε να μας απαντήσετε κυρία Ιβάνοβα έχουν πει πολλά πράγματα. Συναδελφοί μου και εγώ συμμεριζόμουν τα περισσότερα από αυτά, λέει ο κ. Χάβη Λόπε. Θέλω να επισημάνω όμω περισσότερα ω ένα σύστημα. Μιλάμε για 5 εκατομμύρια ανθρώπου. 5 εκατομμύρια νέων στην Ευρώπη που σήμερα δεν έχουν θέση εργασία. Και το 22% της ανεργίας είναι το ποσοστό της ανεργίας των νέων, αλλά αυτό εξαρτάται πάρα πολύ. Είναι 50% στην ε, ε, Ισπανία, αλλά 8% μονάχα στη Γερμανία. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ομοιόμορφες στατιστικές για τα θέματα. Η έκθεση σας είναι πολύ καλή, είναι πλήρη, είναι απαραίτητη, είναι χρήσιμη, όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, γιατί θέλουμε να επικρίνουμε και να θέσουμε εμπόδια στην προσπάθεια που γίνεται, όχι επειδή θέλουμε να καθυστερήσουμε την εφαρμογή τη εγγύηση για του νέου. Καθ' άλλο θεωρούμε ότι είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Πρέπει να είναι χρήσιμη λοιπόν αυτή η εγγύηση. Αυτά τα οποία ελέγχθηκαν, τα οποία τα είχαμε ήδη διαπιστώσει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τα είχαμε ήδη αρχίσει να τα διαβλέπουμε. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε τη συνολική εκτίμηση που να είναι αξιόπιστη για το πόσοι πόροι θα είναι απαραίτητοι για να ευδοκιμήσει αυτή η εγγύηση για τους νέους για να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι αυτή της εγγύησης για των νέων. Δεν έχουμε κριτήρια σε σχέση με το τι είναι η απασχόληση ποιότητος και ο στόχος μας δεν είναι απλώς να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόληση, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόληση με ποιότητα και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να συμφωνήσουμε για το τι είναι η ποιότητα και πώς μπορούμε να ασκήσουμε μια δημόσια πολιτική. Χωρίς κάτι τέτοιο θα δημιουργήσουμε νέες μορφές επισφαλούς εργασία. και αυτό δεν πρέπει να είναι ο στόχος μας των πολιτικών που θέλουμε να ασκήσουμε. Τρίτον, είναι γεγονός ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν ένα μέλλον μεγάλο μέρο τη ότι μπορούμε να μάθουμε αμοιβαία από τι εμπειρίε των κρατών μελών. Αλλά σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι τα κράτη μεταφέρουν τα προβλήματά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για ορισμένα ευρωπαϊκά προγράμματα τα κράτη-μέλη δεν κάνουν τα απαραίτητα για να τα εφαρμόσουν. Δεν έχει να κάνει με θέματα κομματικού χαρακτήρα μονάχα, αλλά υπάρχουν προβλήματα και ελλείψεις στην εφαρμογή των κοινοτικών ενωσιακών προγραμματών. Δεν υπάρχουν ε, αυστηροί μηχανισμοί αξιολόγηση κάτι το οποίο έχει επικριθεί και κάτι τέτοιο απαιτείται πράγματι. Αλλά υπάρχουν μερικά κοινά σημεία, δηλαδή το πρόγραμμα αυτό που αφορά 5 εκατομμύρια νέων. Μας λέει το Ευρωβαρόμετρο γι' αυτό ότι δύο, δύο για κάθε 10 νέους μονάχα ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Μόνο 4% των νέων ξέρουν τι είναι αυτή η εγγύηση για των νέων. Αυτό είναι φυσικά ένα τεράστιο εμπόδιο για την αποτελεσματικότητα του προγράμματο. Ότι δεν γνωρίζουν οι νέοι για το θέμα αυτό. Για να σα δώσω μερικά ακόμα στοιχεία στην Ισπανία. Και σα λέω ότι αυτό ισχύει καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά πιο ειδικά στην Ισπανία έχουμε 800.000 τέτοιους νέους και μόνο 48 χιλιάδες έχουν εγγραφεί σε αυτό το πρόγραμμα. Όχι ότι ε, εποφελούνται από το πρόγραμμα, έχουν εγγραφεί σε ένα κατάλογο, έχουν ζητήσει πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές κτλ. Αυτό όμως σας δείχνει ότι από τους 800.000 μόνο το 6% έχει ασχοληθεί με το πρόγραμμα αυτό. Σας τα λέω αυτά γιατί πίσω από όλα αυτά τα στοιχεία και τα λέω αυτά πάρα πολύ ειλικρινά δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να αρχίσουμε να κάνουμε αντιπολίτευση σε κάποια κυβέρνηση. Υπάρχει μια πραγματικότητα στην Ισπανία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει ελάχιστη γνώση λοιπόν στην Ισπανία για τα θέματα αυτά. Τα νέα στοιχεία από το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο στην Ισπανία που χρησιμοποιεί και το κράτος έλεγαν ότι ένα στα κάθε τρία παιδιά στην Ισπανία είναι φτωχό. Είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. 30% του πληθυσμού ζει σε μια κατάσταση που είναι είτε ε, ένδια είτε κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού. 45% των Ισπανών δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπών. Τα 25% δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν πρόσθετα, πρόσθετες απρόβλεψες να 50 ευρώ. Και πάρα πολλοί δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει η κυβέρνηση. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι σε πολλές χώρες Έχουμε τον ένα στους τρεις να είναι πραγματικά φτωχός και να είναι παιδιά 16-17 χρονών πρέπει να μπουν σε μια εργασιακή αγορά που υπάρχει 50% ανέργεια. Πώς θα μπει αυτό το παιδί στο χώρο εργασίας. Πώς θα θεωρήσει ότι τον καλύπτει το κράτος του, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιοδήποτε άλλος φορές. Αυτό δεν είναι θέμα κόμματος που είναι στην εξουσία. Είναι κάτι που ξεπερνάει τα όρια τα κομματικά και τα όρια της απλής κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ιβάνοβα, πολλοί φόβοι εκφράστηκαν, αλλά και μεγάλη αφοσίωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ αξιότιμοι ευρωβουλευτές για τα πολύ ενδιαφέροντα σχόλιά σας και πρέπει να πω ότι για μας είναι πάρα πολύ πολύτιμο να ακούμε τι μας λέτε κι εσείς, γιατί έτσι μπορούμε να συνεργαστούμε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάθε ερώτηση. Δεν είναι η τελευταία έκθεση που προετοιμάζουμε για την απασχόληση των νέων. Προγραμματίζουμε σειρά εκθέσεων και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε και πάλι την έκθεση ελέγχου για τις ομάδες δράσης για τους νέους. Είναι μια προσπάθεια ε, πιο διεξοδικού ελέγχου για την κατάσταση των νέων σε επίπεδο κράτους μέλους. Είναι λοιπόν η αρχή σήμερα, αλλά όχι το τέλος των προθέσεών μας ε, να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε σε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Πολύ σημαντικά ζητήματα ε, θέσατε σήμερα. Θα αρχίσω, αρχίσω με αυτά ε, που είπε η κυρία Μωρέν Σαρτιέ. Αναφέρθηκε στο θέμα ε, του προγράμματος εγγύηση για την νεολαία ε, έναντι του πρωτοβουλίες για την απασχόληση των νέων είναι ένα κοινό σφάλμα αυτό. Ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει τη διάρκριση μεταξύ των δύο και γι' αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε στην έκθεσή μας να είναι σαφέστατο ε, περί τίνος πρόκειται κάθε φορά να γίνεται μια ε, γρήγορη παρουσίαση των πηγών χρηματοδότησης και ελπίζω να είναι σαφέστερα τώρα όλα, γιατί όπως είπατε κι εσείς η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική για την επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας. Οι νέοι νέοι μας δεν γνωρίζουν, δεν καταλαβαίνουν ε, τι τους προσφέρεται, τότε δεν είναι καμία έκπληξη, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν πηγαίνει κανείς ε, να ε, εγγραφή στις υπηρεσίες αναζήτησης απασχόλησης. Το δεύτερο ερώτημά σας ε, για το θέμα της έλλειψης προγραμμάτων. Με ρωτήσατε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη περισσότερων προγραμμάτων. Η έκθεση αυτή δεν πραγματεύεται το θέμα αυτό, αλλά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή των προγραμμάτων τους, αλλά ε, αν το ερώτημά σας έχει να κάνει με ε, το πρόβλημα των κινδύνων που έχουμε εντοπίσει, είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση δεν υπάρχουν και προγράμματα. Η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης από τα κράτη-μέλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυσχεραίνει το να καταλάβουμε πόσα χρήματα χρειαζόμαστε από την άλλη πλευρά υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν ε, ε, περιορισμούς στον προϋπολογισμό τους. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε που έχουμε μια δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση, που έχουμε περιθώρια και γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επεσήμανε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να θέσουν προτεραιότητες, ποια μέτρα είναι πιο σημαντικά, ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν πρώτα και είναι κάτι το οποίο αναφέρουμε και εμείς στην έκθεσή μας. Ειδικότερα τώρα στο θέμα της, ειδικότερα στο θέμα της δημοσιονομικής, ε, των δημοσιονομικών ε, περικοπών. Είπατε και εσείς ότι σε επίπεδο ένωσης ε, έχουν ληφθεί μέτρα, έχει σημειωθεί πρόοδος, ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έκθεση προχρηματοδότησης και σε επίπεδο επιτροπής. Έχουμε λοιπόν κάνει τη δουλειά μας, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι μια κοινή ε, διαχείριση αυτή της κοινωνικής πολιτικής. Απ' την άλλη κατακράτη κράτη-μέλη που επίσης πρέπει και εκείνα να παίξουν το ρόλο τους. Πολλοί έξιμών και εσείς κυρία Μωρέν Σατιέ αναφερθήκατε στο θέμα της καλής ποιότητας προσφοράς. Είναι πράγματι ένα ουσιαστικό τμήμα της εκθεσής μας ε, για τους κινδύνους και, τις, και για τις συστάσεις μας. Αυτό που εμείς προτείνουμε δεν είναι υποχρεωτικό. Εμείς προσπαθούμε να ε, κάνουμε μια επικοδομητική ανάλυση και να εντοπίσουμε κινδύνους που έχουμε αναγνωρίσει και εμείς. Τα κράτη-μέλη ε, καλούνται ε, σεβόμενα την επικουρικότητα να αποφασίσουν στο πλαίσιο της δικής τους κατάστασης τι μέτρα πρέπει να ακολουθήσουν εμείς. Τα πορίσματά μας τα βασίζουμε σε διάφορα στοιχεία που προέρχονται για παράδειγμα από το πρόγραμμα πλαίσιο ε, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το θέμα της μαθητείας ε, και τις ελάχιστες προδιαγραφές για την άσκηση και τη μαθητεία ε, για να μην υπάρχει, αξιο... να μην υπάρχει εκμετάλλευση των, επιχει... των νέων από τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν επίσης πολλά έγγραφα που θέτουν συγκεκριμένες αρχές σε σχέση με την καλή ποιότητα της προσφοράς Προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε να λάβουμε υπόψη μας και τους δείκτες ε, ε, ποιότητας ε, της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όλος αυτός ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών που κάνουν μία προσφορά να είναι καλή ποιότητα ή όχι, η διάρκεια, το είδος της σύμβασης, ε, αν είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ε, μερικής ή πλήρους απασχόλησης, όλα αυτά βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικές πτυχές, όπως επίσης το επίπεδο προδιαγραφών που απαιτούνται, η διαρκεια το ειδος της συμβασης αν ειναι ορισμενου η αοριστου χρονου μερική η πληρους απασχολησης ολα αυτα βεβαια ειναι παρα πολυ σημαντικες πτυχες οπως επισης το επιπεδο προδιαγραφων που απαιτουνται η σχετικη η ε, εκμάθηση κατά τη διάρκεια της απασχόλησης νέων δεξιοτήτων κλπ. Ε, όλα αυτά βέβαια με πλήρη σεβασμό της επικουρικότητας και για να είμαι και δίκαιη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είναι κάτι το οποίο το είπε και η κυρία Ζούμπερ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε απολύτως τίποτε σε σχέση με τον ορισμό αυτό της καλής ποιότητας πρόσφορας. Κάποια κρατημέλη ε, μετά την καθοδήγηση του Απριλίου του 2014 ε, ε, προς, κάποια κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως αναθεώρησε αυτό το θέμα της καλής ποιότητας προσφοράς, όχι πλήρως βέβαια, δεν ε, κάλυψε δηλαδή διεξοδικά όλα τα χαρακτηριστικά που ανέφερα προηγουμένως, αλλά ούτως ή άλλως και τα κράτη-μέλη πρέπει και εκεί να, να ε, παίξουν το δικό τους ρόλο. Ο κύριος Μπένιφεϊ μας ε, μίλησε για το ρόλο της ε, ανάλυσης ως αντικειμενικής τοποθέτησης, δηλαδή προσπαθούμε να είμαστε ουδέτεροι να μην τοποθετούμε τα πολιτικά σε σχέση με ορισμένες, ε, σε σχέση με το, με το, με το θέμα αυτό που αφορά τους νέους και συμφωνώ απολύτως, έτσι βλέπουμε και εμείς το ρόλο μας. Μιλήσατε για την πολύ ε, κακή κατάσταση στην Ιταλία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σχολιάσω για τα κράτη-μέλη ξεχωριστά, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, αυτή την απάντηση θα μπορέσουμε να σας την ε, παράσχουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει λεπτομερέστερη ανάλυση σε επίπεδο κράτους μέλους. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα πράγματα μόνο ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο από την ε, εγγύηση για την νεολαία, χρειαζόμαστε στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα αναφερθήκατε στην αντίσταση των νέων. Είναι κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με την ε, στρατηγική, την επικοινωνιακή που έθεσε η κυρία Μορέν Σαρτιέ. Και θα ήθελα μία ακόμη φορά να πω την αρχή της κοινή διαχείρισης. Ε, έχουμε την Επιτροπή, έχουμε το Κοινοβούλιο, αλλά έχουμε και τα κρατημέλη, τα οποία και τα κρατημέλη είναι υπεύθυνα για την ε, εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Η κυρία Ζητάνσκα από τη Σλοβακία, κάνατε μια συγκεκριμένη ερώτηση για τα κράτη-μέλη. Να σας παραπέμψω στην, απο... απάντηση που έδωσε και προηγουμένως. Δεν ξέρω σε αυτή τη φάση ποιο κράτος μέλος ε, θα λάβει επίσκεψή μας, γιατί συνήθως 4-5 ε, μέλη επισκεπτόμεθα στο πλαίσιο μίας έκθεσης ε, για να έχουμε μια πιο λεπτομερή εικόνα της κατάστασης. Οπότε για την ώρα δεν μπορώ να μοιραστώ αυτή την πληροφορία μαζί σας, αλλά αυτή τη στιγμή ε, θα είμαστε έτοιμοι. Με πολύ χαρά θα ε, ξαναέρθω και θα σας απαντήσω το θέμα της καλής ποιότητας προσφοράς που θέσατε εσείς. Νομίζω ότι το απάντησα ήδη. Κυρία Ζούμπερ, είπατε ότι η εγγύηση για την νεολαία δεν φαίνεται να είναι πολύ διαφορετική από άλλα μέτρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού ε, Ταμείου. Ναι, είναι γεγονός ότι ξέρουμε κάποια ε, μέτρα ότι έχουν εφαρμοστεί για πολλά χρόνια μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η έλλειψη δεδομένων είναι επίσης ένα θέμα το οποίο και εμείς εντοπίσαμε στην έκθεσή μας. Ε, η έλλειψη δεδομένων ε, είναι ένα τεράστιο κίνδυνο και το αναγνωρίσαμε κι εμεί, Αλλά και πάλι τα δεδομένα αυτά, ε, εδώ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλει να πάρει το λόγο, μπορεί βεβαίως να συμπληρώσει αυτό που, αυτά που λέω εγώ, αλλά δεν μπορούν να παρέχουν δεδομένα αν τα δεδομένα αυτά δεν έχουν προηγουμένως ε, διατεθεί από τα κράτη-μέλη. Αν τα κράτη-μέλη δεν πούν ποιες είναι οι ανάγκε τους. Μιλήσατε επίση και εσείς για την καλή ποιότητα της προσφοράς, νομίζω ότι το κάλυψε και αυτό. Και επίση ρωτήσατε τι θα έπρεπε να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξασφαλίσει ότι αυτές οι συστάσεις ε, εφαρμόζονται. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που ήδη κάνετε. Το ενδιαφέρον και η, αφοσίωση που βλέπω από πλευρά σας σήμερα δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα για σας και δεν νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο ε, βήμα ε, όλης αυτής της σειράς μέτρων που θα ε, λυθούν κατά τη, από τη δική μας την πλευρά είναι απλώς μία πρώτη έκθεση αλλά είμαι βέβαιη ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα που μπορούν να γίνουν. Κυρία Ατζέα και εσείς μας ε, μοιραστήκατε μαζί μας κάτι τρομακτικά νούμερα από τη δική σας χώρα συμφωνώ εγώ μαζί σας απολύτως και με τον κύριο Μπένιφεϊ ότι ε, η εγγύηση δεν αποτελεί πανάκαια. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να συνδυαστεί με πολλά άλλα μέτρα ε, τα οποία ε, πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, προχρηματοδότηση και τα αριθμητικά στοιχεία. Νομίζω ότι μέχρι τον Ιούνιο θα υπάρξει μια έκθεση από τα κράτη-μέλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ε, κονδύλια που έχουν χρησιμοποιηθεί και αυτά που δεν έχουν απορροφηθεί θα έπρεπε να επιστρέψουν στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Τώρα θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. Το παρακολουθούμε εμείς με πολύ προσοχή και θα σας ενημερώσουμε. Κυρία Μάκιντάιρ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Αναφερθήκατε στην ε, μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου ε, πράγματι σημειώσαμε και εμείς ότι δεν εκπονήθηκε μια τέτοια μελέτη στην προκειμένη περίπτωση και πάλι δεν θέλω να πάρω και να έχω πάλι το ρόλο ε, να, να μιλώ εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απλώς να πω ότι ο, ολόκληρη η ιδέα προέκυψε κατεπηγόντως, οπότε ίσως ήταν ένας από τους λόγους ε, αυτό ότι ακριβώς ε, ε, ε, όλα αυτά προέκυψαν ω απάντηση σε μια επίγουσα κατάσταση. Εντάξει, προφανώς αυτό δεν είναι δικαιολογία για την μη διεξαγωγή μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου, αλλά θα το ξαναπώ, χρειαζόμαστε στοιχεία από τα κράτη-μέλη για τις ανάγκες χρηματοδότησης. Αναφέρθηκε στην έκθεσή μας ότι η υποβολή εκθέσεων ε, δεν είχε προβλεφθεί να γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά περιμένω να δω και τι θα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ε, απάντηση σε σχέση με τη συγκεκριμένη υποβολή εκθέσεων. Είναι κάτι το οποίο υπήρχε ως δήλωση, αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι τελικά θα υποβάλει την έκθεση αυτή συμφωνώ ότι η συνεργασία με τα κράτη-μέλη είναι ουσιαστική σημασία, να επικεντρωνόμαστε και στις βελτιστές πρακτικές, όχι μόνο στα αρνητικά αποτελέσματα αυτό. Είναι μια αρχή που προσπαθούμε και εμείς να την ακολουθήσουμε στις ειδικέ μας εκθέσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου, να μην δείχνουμε μόνο αρνητικά παραδείγματα, αλλά μια ε, εξισορροπημένη αντικειμενική θεώρηση των καλών πρακτικών όταν υπάρχουν και όπου υπάρχουν. Κύριε Λόπες, είπατε κι εσείς, μας αναφέρατε κάποια όχι πολύ ευχάριστα αριθμητικά στοιχεία για την ποιότητα των προσφορών. Ναι, αυτό το συζητήσαμε ήδη το θέμα της καλής ποιότητας προσφοράς. Δεν νομίζω ότι η βελτίωση των στατιστικών θα πρέπει να είναι μια απλώς προσωρινή βελτίωση για να δείξουμε ότι κάποιοι νέοι απασχολήθηκαν για κάποιες εβδομάδες και μετά αποχωρούν πάλι από την αγορά εργασίας. Πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο που θα εξασφαλίζει ότι οι νέοι δεν είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης ως ε, ε, φθηνή πηγή ε, εργασίας. ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά αν κάποια θα παρακαλώ να μου το πείτε για να την απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τα είπατε όλα. Ήσασταν πάρα πολύ αποτελεσματικοί και πάρα πολύ πλήρης. Απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα και σε όλες τις ανησυχίες των βουλευτών μας. Νομίζω ότι η έκθεσή σας θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Διότι το θέμα αυτό, το θέμα της ενεργείας των νέων και η πρωτοβουλία απασχόληση των νέων είναι, αν θέλετε, το πιο υψηλού επίπεδου πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή μας. Θα επανέλθουμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Όταν ετοιμαζόμαστε λοιπόν για την αντιμετώπιση της πρότασης Κομισιόν και ενδεχομένω ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και μια παρέμβαση και από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου για το θέμα αυτό θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί η συζήτηση εδώ αφορούσε και αυτά που κάνουν ή που δεν κάνουν τα μέλη κράτη. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Okay, then we'll go to... Και τώρα πάμε στο σημείο 16. Έκθεση για τα αποτελέσματα της εφαρμογής και τη γενική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους για την ενεργογύρανση και την ελληνική των γενιών. Είχαμε κάνει συζήτηση για το θέμα αυτό στο παρελθόν. Αλλά αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε να εξετάσουμε την έκθεση εφαρμογής και συζητήσαμε κύριε Κούκαν το έγγραφο εργασία σας τον Απρίλιο και τώρα μπορείτε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία σε σχέση με την έκθεσή σας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διακεκριμένοι συνάδελφοι κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω λέγον ότι είναι μια μεγάλη τιμή για μένα να παρουσιάσω την πρώτη μου έκθεση, την πρώτη μου από εξανέκαθεν στην Επιτροπή Απασχόλησης και μάλιστα για ένα θέμα το οποίο νομίζω θα είναι ιδιαίτερα προεξάρχον στα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε ήδη από τώρα το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα θέματα γύρανσης και γυρασκότητος. Αυτό βασίζεται μονάχα, όχι μονάχα στα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στην έκθεση της Κομισιόν, αλλά και βασίζεται στο γεγονός ότι τα στοιχεία αυτή θα οδηγήσουν και σε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά. Εξ αρχής λοιπόν, θέλω να πω ότι εδώ έχουμε μία έκθεση για να αξιολογήσουμε το έτος 2012, το γυρεύω αυτό έτος, αλλά η δική μου έκθεση θα προτείνει και κάποιες οδούς για το μέλλον και αντιμετώπιση κάποιων πρακτικών ζητημάτων. Πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω δύο πράγματα σαφή. Η ενεργός γύρανση, όπως την κατανοώ εγώ, δεν είναι ένα εργαλείο για να κρατήσουμε τους ε, ηλικιωμένου για περισσότερο χρόνο στην αγορά εργασίας. Είναι ένας τρόπος να εξασφαλίσουμε υψηλή ποιότητα ζωής, δυνατότητες απασχόλησης για τους ηλικιωμένου και για να άρει διακρίσεις εις βάρος τους. Έτσι βλέπω την ενεργογύρανση και χάρη τα 28 κράτη-μέλη μας και τις μεγάλες διαφορές που έχουν στις πολιτικές αντιμετώπισης της γύρανσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Κάποιες χώρες υπολείπονται ιδιαίτερα και θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να βελτιώσει τη στοχοθέτηση τη χρηματοδότηση για την ενεργό γύρανση. Ο στόχος της έκθεσης αυτής θα ήταν να δώσει μια ρεαλιστική επισκόπηση του Ευρωπαϊκού έτους 2012. Ρεαλιστική λοιπόν προσέγγιση το 2012. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το ευρωπαϊκό αυτό έτος ενεκρίθη καθυστερημένα κάπως και με μικρό προϋπολογισμό. Αυτό δείξε σε καθυστερήσεις αδειρήτως. Πιο σημαντικό όμως είναι να μπορέσουμε να δώσουμε συνέχεια στις πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει κατά και του έτους αυτού και να τις κατευθύνουμε προς την κατεύθυνση μιας στεναρής πολιτικής δέσμευσης. Το θέμα αυτό θα πρέπει να παραμείνει επίκαιρο, όχι μονάχα να αποθνίξει όπως και το έτος 2012. Κάποιοι από τους στόχους του 2012 επετέφθησαν εν μέρη και υπήρξε αυξημένη συνειδητοποίηση Είναι σημαντικό λοιπόν, παραδείγματο να προσαρμόσουμε τον κατάλογο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου για την ενεργή, ενεργό γύρανση που να περιλαμβάνει αρχές για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, τον δίκτυ ενεργού γύρανσης στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημογραφική αλλαγή και να υπάρξει περισσότερη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ δεν δημιουργούνται νέα δίκτυα στον τομέα και ορισμένοι κοινωνικοί εταίροι και ιδιωτικέ επιχειρήσει δεν έχουν ε, υπησέλθει καθόλου στη συζήτηση. Γι' αυτό προτείνω να εντατικοποιήσουμε το τρίγωνο του συντονισμού που βασίζεται στους λήπτες αποφάσεων, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές, την κοινωνία των πολιτών κατά δεύτερον και τον ιδιωτικό τομέα κατά τρίτον. Όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ακόμα διακρίσεις λόγω ηλικίας. Αντιμετωπίζουν στερεότυπα, κλισέ και φράγματα. Στην έκθεση αυτή ζητώ από τα κατημέλη να εφαρμόσουν οδηγία για την ίση αντιμετώπιση με ένα σε ό,τι αφορά την απασχόληση και την εργοδότηση και ζητώ επίσης από την Κομισιόν να αποδώσει την πρέπουσα σημασία στο να αντιμετωπίσει την ανεργία για τους ανθρώπους που είναι πάνω από 50 ετών και επιπλέον θίγω το θέμα της ε, αργυράς οικονομίας ή αργυρά οικονομία, καλύτερα από την κρίζα οικονομία, που δίνει οικονομικές ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν από τον γυράσκοντα πληθυσμό. Κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν ότι εγώ θέλω να πουλήσω στην αγορά τους ολικιωμένους. Όχι, δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσω και παραθέτω ότι πρέπει να έχουμε μια πολιτική η οποία αντιμετωπίζει τι ανάγκε του γυράσκοντος πληθυσμού επί τη βάση τη οικονομική ευκαιρία που θα τους παρέχει και η οποία προκύπτει από τις ε, δαπάνες που μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και που συνδέεται με συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται με την γύρανση και καινοτόμες αντιμετωπίσει για να καλυφθούν οι ανάγκες τους και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέες θέσεις απασχόλησης υπηρεσίες. Οι υπηρεσίε υποστήριξης και μέρημνας θα πρέπει να κατευθυνθούν προς τους καταναλωτές, αυτήν την περίπτωση στους αργυρο, αργυρόμαλους ηλικιωμένους. Τέλος πιστεύω ότι ο εθελοντισμός είναι πολύ σημαντικός και στην ενεργογύρανση και στην διαγενειακή αλληλεγγύη. Κυρία Πρόεδρε, προσβλέπω ιδιαίτερα στο να συνεργαστώ με τους σκιώδεις συζητητέ παρά τη νεότητά του και επίση με οποιοδήποτε άλλο που ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό. Η προθεσμία τροπολογιών είναι η 3η Ιουνίου, Επομένω έχετε ακόμα κάποιε μέρε για να καταθέσετε τροπολογίε και θέλω να πω ότι είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε συζήτηση η οποία μπορεί να γίνει για το θέμα αυτό. Όποιοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται μπορούν να έλθουν να με βρουν. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Thank you. Ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κ. Δησούτε δεν είναι εδώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφο Δικεβιτσούτε δεν ε, μπορεί να έρθει εδώ, ζητά συγγνώμη. Εχθές ε, έκλεισε ξαφνικά το αεροδρόμιο των Βρυξελών και δεν μπορούσε να έρθει και μου ζήτησε να διαβάσω το μήνυμά της. Ευχαριστεί τον εισηγητή για την πολύ καλά προετοιμασμένη έκθεσή του σχετικά με το έτος που αφορά στην ε, διαγενειακή αλληλεγγύη. Η έκθεση εξετάζει τα πιο σημαντικά στοιχεία ε, των ε, κριτηρίων και τα πιο σημαντικά θέματα αυτού του ευρωπαϊκού έτους. Πιστεύει επίσης ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν όλες τις απαραίτητες αξιολογήσεις ε, πριν ε, καταλήξουν για το έτος ε, συνταξιοδότησης να βρουν εργασία όλοι άνω των 50 ε, γιατί με τον τρόπο αυτό δεν θα αυξάνεται η ανεργία. Δεν θα υπάρξει λύση για τα συστήματα κοινωνικής προστασίας της χώρας μας αν δεν ληφθούν υπόψη αυτά τα θέματα. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ότι ε, το γεγονός ότι ε, μόλις τον 12 λήπτει η απόφαση σχετική με τα θέματά μας, αυτό οδήγησε σε καθυστερήσεις. Θα πρέπει λοιπόν ε, να μάθουμε το μάθημά μας για μελλοντικά, για το μέλλον. Τέλος, κύριε κυρία θέλει να στηρίξει την άποψη του εισηγητή ότι ο συντονισμός ανάμεσα στο επίπεδο λήψης αποφάσεων της κοινωνίας των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να ενταθεί, διότι η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού έτους 2012 από την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατέληξε ομόφωνα και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, δεν εκλήξαν σχεδόν καθόλου να συνεργαστούν. Τέλος, η κυρία Βικεβιτσούτα αναφέρει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις καλές πρωτοβουλίες που ελήφθησαν με το έτος το 2012, διότι η γυράσκουσα κοινωνία είναι μια συνεχής απειλή για όλους μας και οφείλουμε να αναζητήσουμε ε, βιώσιμους τρόπους ε, έτσι ώστε να και να το πρόβλημα μακροπρόθεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μου επιτρέψετε, λέει ο κύριος Κρατσνομπεύσκη, ε, να μιλήσω πολωνικά. Γιατί κουράστηκα. Είμαι πολύ κουρασμένος και δεν μπορώ τώρα να μιλήσω αγγλικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ε, πρόταση και την εισήγηση. Αν λοιπόν συγκρίνουμε την Ευρώπη με τις Ηνωμένε Πολιτείε, θα διαπιστώσουμε ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά για τη γύρανση. Δεν έχουμε κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσουμε προκαταλήψεις έναντι των ε, ηλικιωμένων και δεν έχουμε κάνει τίποτα για αυτούς που έχουν αποκλειστεί από την κοινωνία μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δίκαια λοιπόν υποστηρίζεται ότι είναι πολύ σημαντικός ο διάλογος ανάμεσα στις γενναίες και πολύ σημαντική και η επαγγελματική δραστηριότητα των ηλικιωμένων ανθρώπων. Βέβαια, όπως και ο εισηγητής και εγώ και γενικότερα εμείς στην Πολωνία διαφωνούμε να αυξηθεί το έτος συνταξιοδότησης, κυρίως τώρα που έχουμε τόσους πολλούς νέους άνεργους. Κατά την άποψή μου υπάρχουν δύο πράγματα που λείπουν σε αυτήν την έκθεση και ίσως μπορεί κανείς να τα συμπληρώσει μέσω των προστικών. Δηλαδή θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η κατάσταση των ηλικιωμένων ε, ποικίλει στα διάφορα κράτη-μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως όσον αφορά στην ε, σωματική τους κατάσταση. Σε κάποιες χώρες το 70, η ηλικία των 70 δεν λέει τίποτα. Δεν είσαι ηλικιωμένος. Σε άλλες πάλι χώρες Οι άνθρωποι έχουν εργαστεί σκληρά και εκεί η ηλικία των 70 ετών είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Άρα δηλαδή οι κοινωνίες μας ποικίλουν και η κατάσταση και των ε, ηλικιωμένων ποικίλει και αυτή. Εσείς το αναφέρετε λιγάκι αυτό, αλλά όχι επαρκώς. Κατόπιν, ε, στο σημείο υπαριθμών 9 αναφέρεται ότι η ενεργός γύρανση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως ένα μέτρο για να παραμένουν οι άνθρωποι περισσότερο στην αγορά εργασίας. Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι οι ηλικιωμένοι πρέπει να διαδραματίζουν και άλλο ρόλο. Ε, Παραδείγματος χάρη στην οικογενειακή ζωή, στην ε, προαιρετική και εθελοντική εργασία. Αυτό είναι κάτι το σημαντικό στην κοινωνική ζωή και ίσως πρέπει και αυτό να το υπογραμμίσουμε και να πούμε ότι υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί ρόλοι στην κοινωνία. Δεν πρόκειται μόνο για την ε, απασχόληση και την εργασία. Βεβαίω και αυτή επιτρέπει να συμμετέχει κανείς ενεργά στην κοινωνική ζωή. Αυτά από δική μου πλευρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, από τους ε, φιλελεύθερους θα μιλήσω κι εγώ σλοβενικά για να έχουν έτσι και διερμηνείς μας την ευκαιρία να μεταφράσουν από σλοβενικά. Κοιτάξτε, όσον αφορά την ε, συζήτηση που προηγήθηκε, Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του ευρωπαϊκού πληθυσμού, πολλούς Ευρω... Ευρωπαίους δηλαδή. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές χώρες ε, οι οποίες λόγω της οικονομικής κρίσης ε, αντιμετωπίζουν μόνες τα προβλήματά τους και δυστυχώς σε αυτήν την ομάδα των ηλικιωμένων δεν αποδίδεται ιδέουσα σημασία. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε αυτό το θέμα να το εξετάσουμε με μια συγκεκριμένη πρόταση. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το θέμα της αυτονομίας των ηλικιωμένων. Στη Σλοβενία έχουμε κάποια παραδείγματα καλής πρακτικής. Έχουμε παραδείγματα τα οποία είναι γνωστά ε, κυρίως τους οργανισμούς που ασχολούνται με τους ηλικιωμένους. Έχουμε δηλαδή έναν οργανισμό ο οποίος ε, ασχολείται ακριβώς με αυτό, προάγει την αυτονομία των ηλικιωμένων. Ε, η αυτονομία είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι εξής σημαντικό είναι να βοηθά κανείς και τους υπόλοιπους. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι να μπορεί κανείς ε, να ζήσει με καλύτερες συνθήκες και να μπορεί να ε, δώσει, να προσφέρει σημαντικά. Έτσι λοιπόν ε, με τον τρόπο αυτό νομίζω ότι μπορεί κανείς και να δώσει την εντύπωση ότι αναγνωρίζει αυτή τη μορφή εργασίας που προάγει την αυτονομία των ηλικιωμένων. Και έτσι με τον τρόπο αυτό νομίζω ότι οι οργανισμοί αυτοί ε, τραβούν την προσοχή και για το οικονομικό θέματα. Ε, δεν είναι μόνο ο επαγγελματισμός, αυτό που παίζει ρόλο είναι και να καλύπτεται το οικονομικό κόστος. Και κάτι άλλο τώρα, ε, την αναγκαιότητα να ελέγχονται τα οικονομικά ε, των ε, συνταξιωτικών ταμείων. Εάν λοιπόν έχουμε αποφασίσει να διεξάγουμε πιο αυστηρό έλεγχο στις τράπεζες παρά τις αντιδράσεις, νομίζω ότι είναι σωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίζει προδιαγραφές και να επεκτείνει την επιρροή της και όσον αφορά τον έλεγχο των συνταξιδοτικών ταμείων. Γιατί τα συνταξιδοτικά αυτά ταμεία πολλές φορές είναι τα ταμεία εκείνα στα οποία απευθύνεται κανείς ε, και δημιουργεί ε, τρύπες στον προϋπολογισμό. και να αναφερθώ σε αυτό το οποίο εγώ ονομάζω την εναρμόνιση των προσδοκιών και επιθυμιών σε σχέση με την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη ορισμένες φορές περιμένουν υπερβολικά τα άτομα για να μπορούν να τύχουν των υγειονομικών περιθάλψεων και δεν προκάμουν είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να βρούμε μια κοινή προσέγγιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορεί να υπάρξει και μια σύμβαση σε σχέση με την προστασία των ηλικιωμένων ατόμων μια σύμβαση του ΟΙΕ Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ένας αριθμό κρατών που δεν δέχονται τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης δεν καταλαβαίνω και το γιατί, αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουν καλύτερα τους λόγους για τους οποίους αντίστανται. Τέλος, θέλω να φέρω, να επιστήσω την προσοχή σας και μία ασθένεια που βλέπουμε όλο και περισσότερο στους ηλικιωμένους ανθρώπους είναι τρομακτικά τα δεδομένα είναι οι διάφορες μορφές ασθενειών που μου διαφεύγει το όνομά τους αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε μια στρατηγική ευρωπαϊκή που θα μας επιτρέψει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις μορφές άνοιας και πώς θα αντιμετωπίσουμε τα άτομα τα οποία χρειάζονται θεραπεία. Ε? Um, Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθείς η Ζουμπέρ. Εγώ χρειάζομαι πέντε λεπτά διάλειμμα, εάν συμφωνείτε. Για να συνέλθω λέει η πρόεδρος και μετά θα πάρει το λόγο η κυρία Thank you for that. I will now give the floor to Madam Zuber. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζούμπερ. Nós, uh, em relação a este relatório, uh, enfim, temos... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ορισμένες σκέψεις να σας εκθέσω. Κυρίως ενδιαφέρει ο πραγματικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας για την ενεργό γύρανση. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, διότι γυράσκουμε ήδη διδασκόμενοι και είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνει μια εκστρατεία, αλλά όχι μια εκστρατεία η οποία καλύπτεται από την φενάκη της ενεργούς γύρανσης, ώστε να χρησιμοποιηθούν περισσότερο ηλικιωμένοι στο χώρο εργασία, αντίθετα μια εκστρατεία για την υγιή, υγεία γίδανση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη ηλικία συνταξιοδότησης, ότι θέλουμε τα άτομα να είναι υγιή χωρίς αυτό να συνδέεται με την υποχρέωση να εργάζονται. Το 2012 αναφέρθηκε πάρα πολύ το θέμα της ε, βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και ετέθη ιδιαίτερα επιτάπητος το θέμα του να μπορούν οι ηλικιωμένοι να εξακολουθήσουν να εργάζονται. Δεν πρέπει να είναι αυτό όμως το πνεύμα το οποίο θα μας διατρέχει στη συγκεκριμένη συζήτηση. Το θέμα των ηλικιωμένων σήμερα αντιμετωπίζεται περισσότερο υπό την έποψη των δημοσίων υπηρεσιών που θα πρέπει να τους δίδονται οι υγειονομικές υπηρεσίες όπου υπάρχουν πολλές ελλείψεις που όμως θα πρέπει να είναι ένα δικαίωμα για αυτούς. Θα πρέπει να υπάρχουν οι δομές οι οποίες θα τους επιτρέψουν να συμβάλλουν με ίσο επίπεδο στην ε, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, αθλητική ζωή και αυτό εξακολουθεί ένα πρόβλημα για πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ γλυσχρές οι συντάξεις των ηλικιωμένων, κάτι το οποίο εμποδίζει και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Γι' αυτό, κατά την άποψή μας, το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην, ε, στην ε, δυνατότητα να έχουν καλύτερη υγεία οι ηλικιωμένοι και όχι απλώς να έχουμε το στόχο να συνταξιοδοτούνται αργότερα. Αντίθετα θα πρέπει η περίοδος συνταξιοδότησης των ηλικιωμένων να τους εξασφαλίζει μια ε, αξιοπρεπή ζωή ως ανταμοιβή της συνεισφοράς τους στην κοινωνία. Για να επιληθεί λοιπόν το πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλειας και των, της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικών παροχών πρέπει να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη ανακατανομή του πλούτου και την μεταφορά της υπεραξίας στον τομέα του, των δημοσίων αγαθών και την ε, διανομή της στους πλέον ηλικιωμένους και τους συνταξιοδοτημένους. Η κεφαλαιοποίηση λοιπόν των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας έχει οδηγήσει σε μια υπερσυγκέντρωση του πλούτου και έχει οδηγήσει πολλά άτομα στο να είναι υποχρεωμένα να δουλεύουν στο διηνεκές χωρίς να μπορούν να ζήσουν από τη σύνταξή τους. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι μια υποχώρηση της κοινωνικής προόδου σε όλα τα επίπεδα. Αυτές είναι λοιπόν οι βασικές ιδέες που θα θέλαμε να αναφέρουμε σε σχέση με την έκθεση και κατά τα άλλα συμφωνούμε με πολλές από τις παραγράφους του κυρίου Κούκαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Ζανούκα από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ Και εμείς γνωρίζουμε τη σημασία που θα έχει το κείμενο αυτό για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους για την ενεργό ε, γύρανση. Η δική μου χώρα είναι μία από τις φτωχότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και και μαζί με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία είναι, ε, είναι από τις ε, χώρες τις οποίες τα επίπεδα της συνταξιοδότησης είναι τα χειρότερα. Μας είπε και ο κύριος Κούκαν, ενεργός γύρανση δεν σημαίνει μόνο καλύτερες ε, προϋποθέσεις ε, στην εργασία για τους ε, ηλικιωμένους. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να συμφωνηθεί μεταξύ εισηγητών και σκιωδών εισηγητών. Κάτι που μου προκαλεί έκπληξη είναι ότι πρέπει να υποστηρίξουμε όλους, όλους τους πολίτες στην προσπάθειά τους να ζουν αυτόνομα. Εγώ το βρίσκω λίγο αντιφατικό αυτό, μπορεί να διαφωνεί ο κύριος Κούκαν. Όλοι δηλαδή πρέπει να, ε, να δουλεύουν περισσότερο για να μπορέσουν να ζουν ε, ε, αυτόνομα. Μου φαίνεται λίγο αντιφατικό αυτό επίσης. Μας δώσατε πέντε παραδείγματα προγραμμάτων και μας λέτε ότι δεν είναι διεξοδικός ο κατάλογος. Το ερώτημά μου είναι η Εστονία, η Σλοβακία, η Τσεχία και η Σλοβενία μόνο ε, σε αυτές τις χώρες περιορίζετε τα παραδείγματά σας. Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι πότε πρέπει να υποβάλουμε τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Η Λάουρα Άγκαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον ε, συγητή για όλα αυτά που μας ε, είπε. Τον ευχαριστώ πολύ για το έγγραφο και την εισήγηση παρουσίας, που σε μεγάλο βαθμό ε, συμφωνούμε. Νομίζω λοιπόν ότι γίνεται έτσι λίγο μια οριζόντια τοποθέτηση και ίσως αυτό πράγματι να προσθέσει αξία και στην σύνταξη του τελικού εγγράφου. Η ενεργός γύρανση ε, προφανώς και είναι αξία, συμφωνούμε απόλυτα, είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Είναι πολύ καλό να υπάρχει κοινωνική συμπερίληψη, πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και για άτομα τα οποία είναι πιο προχωρημένα από τους άλλους. Και έτσι θα υπάρξει και γενικότερα κοινωνική συμπερίληψη. Προφανώς ε, και δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, θετική διακριτική μεταχείριση για ορισμένες θέσεις απασχόλησης υπέρ των νέων, ε, γιατί υπάρχουν κάποιοι ηλικιωμένοι ηλικία 55-60 ετών που έχουν βγει από την αγορά εργασίας και δεν τους προσφέρεται η δυνατότητα να επανέλθουν. Κάτι άλλο όπου μπορούμε να έχουμε θετική στάση δηλαδή οι πολιτικές ε, υπέρ της ενεργού γύρανσης ε, δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένα εργαλείο για να ε, διατηρούνται οι άνθρωποι στον χώρο της εργασίας. Εκείνο που πιστεύω είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τάστε κανείς υπέρ του να υπάρχει τέτοιο όριο συνταξιοδότησης που θα επιτρέπει να υπάρχει μια ποιοτική μετάβαση ιδιαίτερα ποιοτική μετάβαση στην ηλικία συνταξιοδότηση. Εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ένας εξ αυτών είναι η διαφοροποίηση των ε, επαγγελμάτων. Γιατί αν παραδείγματο χάρη έχει κάνει κανείς μια βαριά εργασία, ε, δεν είναι το ίδιο και δεν είναι και ίδια η ηλικία αξιοδότηση από το να έχει κάνει κανείς μια καθιστική εργασία. Γι' αυτό λοιπόν Ας μην ε, προσπαθούμε να πούμε ότι η μόνη πολιτική είναι να παρατείνεται η απασχόληση. Θα πρέπει λοιπόν αποφασιστικά να αντιμετωπίσουμε το θέμα των άνω των 50 χωρίς εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εξευρεθούν αποτελεσματικά εργαλεία για να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, για να επανενταχθούν ε, σε νέες τεχνολογίες. Αυτό νομίζω επίσης είναι κάτι το σημαντικό. Και τέλος, ε, η χρηματοδότηση προγραμμάτων που προάγουν την ενεργογύρανση, αυτά όλα θα πρέπει ε, να προωθηθούν όπως και η χρηματοδότηση από ε, διαρθρωτικά ταμεία. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε υπάρχει για να έχουμε μια πραγματικά ποιοτική γύρανση. Επίσης ε, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε λιγάκι και αυτό το νέο χρηματοδοτικό μέσο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ενεργού γύρανσης. Ε, θεωρώ όμως ότι προηγουμένως είναι απαραίτητο να γίνει μια ad hoc μελέτη για να εντοπίσουμε ε, με ποιο τρόπο και ποια κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και τέλος, νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα είδος ε, ένταξης, να υπάρχει ένα πλησίασμα των παλαιών και των νέων γενεών να υπάρχει δηλαδή ένα είδος ε, συμβίωσης ε, διότι πιστεύω ότι βλέποντας ε, σε προοπτική τις διάφορες γενιές νομίζω ότι η μία μπορεί να ωφελήσει την άλλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όπως καρακοί συνάδελφοι την, ε, τοσία σχέδιο που μας έχει παρουσιάσει ο κύριος Κούκαν και το έγγραφο εργασία του και τα δύο έγγραφα είναι πάρα πολύ σημαντικά και αποτελούν μια στερεά βάση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ενώπιον μια κατάσταση η οποία δυστυχώ είναι πολύ δύσκολη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν πιστεύουμε ότι η δημογραφική γύρανση δεν είναι πρόβλημα, 37,5 ήταν ο μέσος όρος του 1992 και το 2050 ο μέσος όρος ηλικίας προβλέπεται να έχει ξεπεράσει τα 50 έτη η μέση ηλικία. Αυτό δείχνει ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Βλέπουμε χώρες όπως είναι η Ισπανία, όπου υπάρχουν περιοχές όπου το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα οξύ. Αν θέλουμε λοιπόν να είναι βιώσιμο το οικονομικό μας και οικονομικό μας μοντέλο, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή γύρανσης στο ταχύτερο δυνατόν χάρη στο Ευρωπαϊκό Έτος Γέρανσης, έχει αυξηθεί η συνειδητοποίηση για την γύρανση του πληθυσμού και για τις δημογραφικές αλλαγές. Σε επίπεδο διάγνωση τα έχουμε πάει πολύ καλά, έχουμε κάνει μια πολύ καλή αξιολόγηση, αλλά συμφωνώ και με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο. Πρέπει να στρέψουμε τα μάτια μας προς το μέλλον και να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να σε θέση να ζήσουν ανεξάρτητα, να εργάζονται εάν το θέλουν μετά από την ηλικία της συνταξιοδότησης και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες συναδέλφους ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους εργαζόμενους άνω των 50 ετών να μπορούν να ζουν σε ένα περιβάλλον διαρκούς μάθησης ώστε να μην είναι αντικείμενο διακρίσεων για λόγους ηλικίας. Όλα αυτά όμως δεν σημαίνουν ότι πρέπει να έχουμε μια ενεργή γύρανση με τον εργάζομαστε αενάγως. Πιστεύω ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί φυσικά η ηλικία συνταξιοδότησης και να προσαρμοστεί στο προσδόκιμο ζωής. Αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία συνάπτονται με την ηλικία, να υπάρχει καλύτερη συμμετοχή στην κοινωνία, μια αύξηση της ποιότητας ζωής και εν τέλει θα ήθελα να σταθώ σε ένα θέμα το οποίο εμένα με ανησυχεί και με απασχολεί ιδιαίτερα έχει να κάνει με τις περιοχές της υπαίθρου, τις περιοχές αυτές που υπάρχουν μειονεκτήματα γεωγραφικά και δημογραφικά, περιοχές που υπάρχει μικρή πυκνότητα πληθυσμού, περιοχές νησιώτικες ή υπηρετικές. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν το πρόβλημα της γύρανσης αλλά συγχρόνως και της απερίμονης σε σχέση με τον πληθυσμό και η έκθεση θα πρέπει ίσως να εστιάσει λίγο περισσότερο στο θέμα αυτό. Στις περιοχές αυτές οι νέοι πολλές φορές πρέπει να φύγουν. Δεν έχουν καμία δυνατότητα να βρουν θέση εργασίας. Επομένως, η δημογραφική γύρανση γίνεται με επιταχυνόμενο και δραματικό τρόπο. Χωρίς νέους δεν υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν υγειονομικές υπηρεσίε. Γι' αυτό θα πρέπει να εργαστούμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Αυτά ήθελα από κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Η προθεσμία κατάσταση των τροπολογιών είναι η 7 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι και η εξέταση των τροπολογιών θα λάβει χώρα στις 23 Ιουνίου η έγκριση στην Επιτροπή Απασχόλησης 15 με 16 Ιουλίου. Περνάμε στο σημείο 17 της ημερήσιας διάταξης το Ευρωπαϊκό τα ευρωπαϊκά Διαφορετικά ταμεία υγιής, οικονομική διακυβέρνηση, Καθεδρία γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο γνωμοδότηση. και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή τον Χάβι Λόπε. Ευχαριστώ πολύ να κάνω μια σύντομη εισαγωγική παρέμβαση για το θέμα το οποίο μας απασχολεί. Έχει να κάνει με την μακρό ερεσιμότητα. Ξέρετε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θεώρησαν ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινή βάση για τον κανονισμό αυτό και όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε που αφορούν τα διαρθωτικά ταμεία ή τα ταμεία επενδύσεων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο οικονομική διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι τώρα μια πραγματικότητα όπω γνωρίζετε πολύ καλά το six pack, το two pack κτλ δίπτυχο, εξάπτυχο και μια σειρά από ειδικέ κατά χώρα συστάσει. Η βασική διατρέχουσα ιδέα ήταν τότε με στόχο την ορθολογικοποίηση τη ε, διοίκηση των Ταμείων Επενδύσεων και διαχωριστικών Ταμείων ήταν να συνδεθεί η δυνατότητα χρήση των Ταμείων αυτών με την μακροαιρεσιμότητα που τότε ήταν υποχάραξη και τώρα εφαρμόζεται οικονομικός, ε, χρηματοοικονομικός και δημοσιονομικός έλεγχος των κρατών μελών. Τότε μια μεγάλη πλειοψηφία από τις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησαν ότι αυτή η σύνδεση που μπορεί να φτάσει μέχρι το σημείο να αναστέλλεται η χρήση των κοινοτικών πόρων σε ένα κράτος γιατί δεν τηρεί τις υποχρεώσεις μακροαιρεσιμότητος στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει με τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι και αντιπαραγωγικό. Και είχαμε καταθέσει και μια τροπολογία στο άρθρο 23 που ήταν τότε άρθρο 21 στο πρώτο έγγραφο για τις κοινέ διατάξεις του κανονισμού. Ε, υπήρξε μια τροπολογία λοιπόν του Αραμκόσακ από το ΕΛΚ που θεώρησε ότι δεν είχε νόημα να έχουμε μια τόσο μεγάλη ερασιμότητα που μπορούσε να οδηγήσει στην αναστολή της δαπάνης των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είχε αυτή την άποψη, γιατί τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν στόχους μακροπρόθεσμους και είναι δύσκολο και προβληματικό να τα συνδέσουμε τα ταμεία αυτά με κάτι το οποίο είναι τόσο συγκυριακό όσο είναι η διαδικασία Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και αυτό μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό γιατί είναι φανερό κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται στη χειρότερη οικονομική κατάσταση σε ό,τι αφορά τι μακροοικονομικέ ισορροπίε είναι αυτά τα οποία πρέπει να καταβάλουν ακόμα μεγαλύτερε προσπάθειε προ την κατεύθυνση αυτή και όμω παρόλα αυτά έχουν περισσότερη ερεσιμότητα να ικανοποιήσουν, επομένω είναι πολύ πιο δύσκολο να μπορέσουν να αποκομίσουν το όφελο από τα διαφορετικά ταμεία που τα χρειάζονται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κράτο. Για όλου αυτού του λόγου, λοιπόν υπήρχε η αμφιβολία που είχε διατυπωθεί και ορθά λέγω σε σχέση με τη δυνατότητα επαναπρογραμματισμού ή αναστολή των διαφορετικών πόρων. Και επίση, ανεξάρτητα από το αν πιστεύει κανεί ότι αυτό δεν έχει νόημα ή ότι είναι αντιπαραγωγικό, αυτό στρέφεται κατά τη ίδια τη φύση των πόρων διάρθρωσης και επένδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν σαν στόχο να προωθήσουν την οικονομική και κοινωνική σύγκληση όλων των καθών μελών και όλων των περιφερειών. του λεχθέντο από τη στιγμή που έχει εγκριθεί αυτό ο κανονισμός και με το ΑΒ23 με τη μορφή που έχει σήμερα, με κάποιες μορφές αιρεσιμότητας που περιλαμβάνονται μέσα στη μακροεκονομική ερεσιμότητα που αναφέρεται στο άρθρο 23, έχουμε αυτή την ε, ανακοίνωση της Κομισιόν η οποία έχει σαν στόχο να συγκεκριμενοποιήσει τις μορφές μη τήρησης της και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αποτιμάται αυτή η μακροαιρεσιμότητα, με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει ο αναπρογραμματισμός σε λειτουργικό επίπεδο των κονδυλίων αυτών ή της αναστολής πληρωμών για τα διαφορετικά ταμεία. Προς την κατεύθυνση αυτή, η πρόταση γνωμοδότησης που κάνω και φυσικά είμαι ανοιχτός να ακούσω τις διάφορες απόψεις που μπορούν να έχουν οι συνάδελφοί μου στην Επιτροπή Απασχόληση και να συζητήσω μαζί τους, όπως ε, είχα κάνει και στην προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρότασή μου σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν να πω πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να εξάρουμε ιδιαίτερα ως Επιτροπή Απασχόλησης το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει στην ανακοίνωσή της ότι τα πολυετή προγράμματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, ιδίως σε μια εποχή αβεβαιότητας και κρίσης, απαιτούν μια σταθερότητα και μια βεβαιότητα και πρέπει να αποφευχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ή ο επαναπρογραμματισμός και να ε, προωθηθεί η σταθερότητα προς όφελος των προγραμμάτων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λέει και η ανακοίνωση της Κομισιόν και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Δεύτερον, θα πρέπει να τονίσουμε ότι μπορεί να υπάρξει έλλειψη συνάφειας και ασυνέχεια και ασυναρτησία όταν αντιμετωπίσουμε σημαντικά ε, ασυμμετρικά σοκ και κλειδονισμού στα κράτη-μέλη και τη στιγμή που ο στόχος πρέπει να είναι η οικονομική και η κοινωνική σύγκληση, δεν έχει νόημα. Είναι ασυναρτησία τα κονδύλια αυτά να μην πάνε σε χώρες οι οποίες είναι αυτές που τα χρειάζονται πολύ περισσότερο από τις άλλες. Αυτό στρέφεται κατά της φύσης αυτών των ταμείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, είμαι ιδιαίτερα προσεκτικό σε σχέση με τους συνολικούς στόχους των κοινών διατάξεων του κανονισμού αυτού που έχουν να κάνουν με τον κοινωνικό χώρο, με την απασχόληση, γιατί με την διαδικασία επαναπρογραμματισμού, εάν εφαρμοστεί το άρθρο 23, μπορούμε να αναστείλουμε χρηματοδοτήσεις και έτσι να επιδεινώσουμε το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας. Τέταρτον, θεωρώ στη γνωμοδότησή μου ότι το άρθρο 23 προφανώς προβλέπει και κάποιες εξαιρέσεις στην εφαρμογή του για χώρες όπου είναι οι πιο σοβαρές οικονομικές συνθήκες σε ό,τι αφορά την ένδια, την ανεργία, την έλλειψη ανάπτυξης και πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να ενισχύσουμε τις εξαιρέσεις αυτές στο άρθρο 63 και ότι, να τονίσω ότι αυτό θα, θα ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη εάν τίθεται το θέμα του επαναπρογραμματισμού των κονδυλίων. Και για να κλείσω, η ανακοίνωση λέει ότι πρέπει να ληφθεί μια απόφαση στο θέμα αυτό και φυσικά η δική μας θέση είναι ότι και το Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφέρουν τη γνώμη τους στην περίπτωση που λαμβάνεται μια απόφαση σε σχέση με το άρθρο 23 και ελπίζω ότι με τους συναδέλφους στα πλαίσια της συζήτησης θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση για τα θέματα αυτά. Κασεντεύσκη, TCR. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θέλω να πω ότι συμφωνώ με αυτά τα οποία λες ε, στην εκθεσή σου. Πράγματι είναι αλήθεια ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς ε, πώς συνδέονται οι μακροοικονομικοί δείκτες, παραδείγματος χάρη με την πολιτική συνοχής. Σήμερα στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε μία διαφορά ανάμεσα στην πολιτική της κυβέρνησης και τα ταμεία. Αυτό μας συμβαίνει στην ε, Πολωνία. Και κάτι άλλο. Ε, μιλήσατε ε, για αυτή την διακοπή των ε, πληρωμών από το Ταμείο Συνοχής. Αυτό ήταν ε, το 2012 και έγινε μόνο έναντι της Ουγγαρίας, ενώ υπήρχαν και άλλες χώρες που δεν τήρησαν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Πολύ σωστά επισημαίνεται ότι ο στόχος ε, αυτών των ταμείων είναι διαφορετικός και ότι τέτοιου είδου εργαλεία οδηγούν σε όξυνση των διαφορών ανάμεσα στις ε, περιφέρειες, κυρίως όταν πρόκειται για χώρες που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Αυτά προς το παρόν και μετά θα σκεφτούμε να δούμε ε, το ποια ακριβώς είναι η τάση διότι αυτό το οποίο ε, έχει σχέση με το άρθρο 23 δεν ξέρω, εγώ το βρίσκω τελείως διαφορετικό. Συγγνώμη που άργησα, περίμενα να τελειώσει η διερμηνία. Εκ μέρου ε, του σκιώδου συζητητή των φιλελεύθερων θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που ε, η οικονομική διακυβέρνηση συνδέεται με τα Ευρωπαϊκά Διευθυντικά Ταμεία ως προς την εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων και ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει μια σημαντική, μια πολύτιμη ε, συμμετοχή ε, η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, οι επενδύσεις να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο κοινωνικό-οικονομικό για να μπορέσουν να μεγιστοποιήσουν ε, την, το, δυναμικό, ειδικότερα, το δυναμικό τους ειδικότερα σε μειονεκτούσες περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προβεί σε ειδικέ αναχώρασεις στάσεις Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πολύ προσεκτικοί όταν θα κληθούν να εφαρμόσουν τα προγράμματα όπως προβλέπεται από τους ε, από τον κανονισμό, ειδικότερα όταν δεν έχουν καταφέρει να προδούβουν σε διορθώσεις τα κράτη-μέλη κατά την εφαρμογή. Ε, οι πολίτες δεν πρέπει να είναι ε, τα πρώτα θύματα της κακής εφαρμογής και είναι κρίμα που οι κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν παραγνωριστεί. Πρέπει να εξασφαλιστεί η δημοκρατική λογοδοσία και η διαφάνεια. Η γραμμή των τροπολογιών που ο σκιώδης εισηγητής μας θα υποβάλει θα είναι να εξασφαλίσει ότι η αναστολή των πληρωμών χρησιμοποιείται ως ε, τελική λύση γιατί η αναστολή των πληρωμών μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο για τις ε, ε, ενδιαφερόμενες περιφέρειες και ειδικότερα αυτές με υψηλό ποσοστό ανεργίας όπως αναφέρεται στο παράρτημα 3 ε, των κοινών διδάξεων του κανονισμού. Ε, πρέπει να ενισχύσουμε την απασχόληση και να προσπαθήσουμε να αντισταθμίσουμε ανεπιθύμητα αποτελέσματα και όταν γίνεται νέος προγραμματισμός ε, της χρηματοδότησης πρέπει να ληφθεί υπόψη το δυναμικό της ε, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της ανάπτυξης και στο πλαίσιο των ειδικών αναχώρας συστάσεων. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Ζούμπερ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα. Πρόκειται για μια συζήτηση που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ήταν πάρα πολύ εύκολη η συζήτηση αυτού του θέματος στο Κοινοβούλιο, ειδικότερα όταν, μιλάμε, όταν βλέπουμε τις προοπτικές για τα διαρθρωτικά ταμεία. Ε, νομίζω, δεν ξέρω κατά πόσο έχει εγκρίνει κάτι τέτοιο η Επιτροπή Απασχόλησης, πάντως Το πρόβλημα είναι ότι πράγματι είναι διαφορετική η δρόμη που ακολουθούμε στην περίπτωση αυτή. Εάν θεωρήσουμε ότι κάτι είναι αντιπαραγωγικό όπως ελέγχθη, αυτό είναι σαφές ότι οδηγεί στον παραλογισμό και αντίκειται προς την ανάγκη αποτελεσματικής χρήσης των ταμείων των ενωσιακών για να μειωθεί η ανισότητα. Εμείς θεωρούμε ότι η αρχή της μακροαιρεσιμότητος από αυτή την άποψη έχει προβληματικό χαρακτήρα. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει ακόμα πια σήμερα μια πλειοψηφία που να υποστηρίζει την αρχή της ε, μακροερεσιμότητος ή το αντίθετο. Και υπάρχουν δύο ή τρεις λόγοι για τους οποίους εμείς θεωρούμε ότι αυτή η αρχή θα πρέπει να ανακληθεί, η αρχή της μοτρονεσιμότητας. Όταν έχουν προσχωρήσει οι χώρες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δυνατότητες των κοινοτικών ταμείων και της διανομής τους δεν είχε καμία απολύτως σχέση με αυτόν τον εκβιασμό που γίνεται με την χρήση της αρχής της μακρορεσιμότητας. Επομένως, οι χώρες είχαν τότε ένα περιθώριο ελιγμών για να αποφασίσουν για το δικό τους μοντέλο ανάπτυξη και το μοντέλο επενδύσεών τους. Αλλά αυτό τώρα αναιρείται. Επίσης όμως και σε σχέση με τις ίδιες αρχές που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν οι πόροι οι ευρωπαϊκοί τις περισσότερες φορές δεν καταφέρνουν να ικανοποιήσουν τους στόχους οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Εγώ δεν μπορώ λοιπόν να κατανοήσω πώς θα πρέπει να προσδέσουμε τους διαχρονικούς πόρους σε τέτοιες ε, συστάσεις που έχουν να κάνουν με την μακροασιμότητα. Εμείς έχουμε μπει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου λόγω της δράσης της Τρόικας. Ακολουθήσαμε φυσικά τις επιταγές της Τρόικας, αλλά η Τρόικα μέσα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μας είπε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε όλες τις συστάσεις της ε, ε, Τρόικα να μειώσουμε το δημόσιο χρέος, κάτι το οποίο σήμαινε να επιδεινώσουμε ακόμα περισσότερο με μέτρα τα οποία περίεστελαν τις δαπάνες, όλα αυτά τα οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι διαδοτικοί πόροι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βοηθούν τα κράτη-μέλη στο να επενδύουν σε πολιτικές που έχουν εναλλακτικό χαρακτήρα που θεωρούν τα κρατημέλη ότι μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση και η περαιτέρω χρήση της μακροερεσιμότητας δημιουργώντας περαιτέρω φραγμούς και εμπόδια, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι αποτελεσματικό. Ο δρόμος του μέλλοντος θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να αποφευχθούν οι αναστολές της χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά ταμεία θα πρέπει να κατανοηθεί ότι είναι κάτι το αντιπαραγωγικό για τα φτωχότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να μην εφαρμόζεται η δυνατότητα της αναστολής με τον τρόπο με τον οποίο είχε καταρχήν υπόψη της η Κομισιόν. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή θα υποστηρίξουμε λοιπόν την γραμμή αυτή οι οποίες καταδικάσουν ουσιαστικά την έννοια της μακροαιρεσιμότητας. δεν είναι Η κυρία Ντέλη δεν είναι εδώ. Είναι κανείς που την εκπροσωπεί. Όχι. Λάουρα Άγγεα. Grazie ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, τη συνάδελφο και βεβαίως ε, τη διαβεβαιώνουμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε. Θέλω να σας πω ότι η χρήση αυτών των κονδυλίων για να βελτιωθεί η οικονομική διακυβέρνηση νομίζω ότι δεν ισχύουν για την περιφερειακή ανάπτυξη και για την κοινωνική ψυχή, διότι ο καθοριστικός τους ρόλος είναι να ενισχύσουν τις κοινωνικές πολιτικές και την εδαφική πολιτική, όπως επίσης και να περιορίσουν τις οικονομικές διαφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν το να ανασταλούν τα κονδύλια, αυτό ενδεχομένω να επιδεινώσει την οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Κυρίω ε, στι χώρε εκείνε, οι οποίε αντιμετωπίζουν πολλέ δυσκολίε λόγω τη κρίση και διότι ε, οι τοπικές υπηρεσίες ε, κινδυνεύουν να κάνουν τελικά λιγότερες επενδύσεις. Είναι λοιπόν απαραίτητο να επιμείνουμε στο να διατηρηθούν αυτά τα κονδύλια και ξεχωριστά από τα άλλα γιατί είναι χρηστή οικονομική διακυβέρνηση. Σας επισημαίνω, δεν θα πρέπει οι περιφέρειες να τιμωρούνται για διάφορα σφάλματα που έχουν γίνει και κυρίως όταν ε, τα σφάλματα αποδίδονται στις ε, εθνικές ε, διοικήσεις. Μην ξεχνάτε κάθε φορά που τιμωρούμε την τοπική αυτοδιοίκηση, κατ' ουσίαν τιμωρούμε, με τιμωρούμε τους πολίτες ε, γιατί αυτοί υποφέρουν και δεν υποφέρει τελικά η διοίκηση. Άρα δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας ε, και εμείς τις δικές μας τις ε, τροπολογίες θα τις καταθέσουμε και θα τα πούμε μεταξύ μας και οι σκιώδεις εισηγητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι Δευτέρα Ιουνίου το μεσημέρι. Α, έγκριση στην Επιτροπή Απασχόληση 23 Ιουνίου, έγκριση στην Επιτροπή RMG 13 με 14 Ιουλίου. Περνάμε το σημείο 18 στην ημέρια διάταξη κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλεις των κρατών μελών είναι η εξέταση 217 τροπολογιών στην έκθεση της κυρίας Αγέας επί τη βάση μιας νομοθετικής πρότασης για απόφαση από το Συμβούλιο για τις κατευθυντήριες γραμμές η έκθεση περιλαμβάνει 29 τροπολογίες. Πήρω το λόγο στην κυρία Αγκαία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους ε, σκιώδεις ε, εισηγητές, τους συναντέλφους που με βοήθησαν στο να συντάξω αυτό το έγγραφο. Διότι Εκείνο το οποίο καθίσταται σαφές είναι ότι παρότι υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις και σημείο κίνησης, υπάρχει βούληση για συνεργασία. Όπως είπε και η Πρόεδρος, κατατέθηκαν πάρα πολλές τροπολογίες. Όμως κατορθώσαμε να επιτύχουμε μια καλή βάση συμβιβασμού. Ε, τι συζητήσαμε στις δύο συναντήσεις και οδών ε, εισηγητών που είχαμε και πέρα από τις διαφορές που ενδεχομένω να υφίστανται για κάποια επιμέρους θέματα, εξακολουθεί να παραμένει ουσιαστικά η δήλωση, η επιτιμία μάλλον, να καταλήξουμε σε ένα ε, έγγραφο με ουσία που θα μπορεί να περάσει στο Συμβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι οι συνάδελφοι έχουν αυτή την καλή θέληση να συνεργαστούν και το ίδιο ισχύει βεβαίω και για τους και Όσον αφορά τους ε, συμβιβασμούς, νομίζω αυτοί αντικατοπτρίζουν το ότι όλοι επιθυμούμε να καταλήξουμε σε μία λύση, να συμβιβαστούμε και βεβαίως ε, ο καθένας ε, αν δεν μπορεί να συμβαστεί, προφανώς και διατηρεί τη δική του τη θέση. Εκείνο που έχει σημασία είναι να υπάρχει ένα ουσιαστικό έγγραφο. Αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν μας ικανοποίησε και αυτό που όλοι λένε είναι ότι θα πρέπει, όπως συνέβη και σήμερα το πρωί, εναντί της Επιτρόπου της κυρίας Τίσεν, οφείλουμε να πούμε ότι είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί τόσο η στρατηγική 2000, να αναθεωρηθεί η στρατηγική 2020, αλλά να παραμείνουν οι βασικοί πυλώνες που είναι η ουσιαστική μείωση της ανεργίας, οι ε, δικλείδες κοινωνικής προστασίας. Με αυτή την προσέγγιση θα ε, προσπαθήσουμε στις κατευθυντήριες γραμμές να αναδιατυπώσουμε τη στρατηγική 2020. Παράλληλα θα προσπαθήσουμε να παραμείνουμε πιστοί στους στόχους μας. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουμε αναλύσει δύο κατευθυντήριες γραμμές και αναδιατυπώνουμε μια καινούργια πρόταση με την συνεργασία των συναντέλφων και με την πολύ καλή δουλειά βέβαια που έχει κάνει η γραμματεία. Μας έχει στηρίξει πάρα πολύ και νομίζω ότι τελικά θα καταρτάσουμε να καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό έγγραφο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος, ο από το Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Λάουρα Αγκαία και νομίζω ότι έχει βοηθήσει ιδιαίτερα και τους σκιώδεις εισηγητές με την αντιμετώπιση που είχε για το θέμα αυτό προσπάθησε να έχει συζητήσεις και συνεργασία μαζί με όλους τους σκιώδεις εισηγητές και γι' αυτό η τόσο σημαντική αυτή έκθεση έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό θέλει να υπάρξει η απαραίτητη απήχηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πνεύμα αυτό το θετικό ήταν φανερό στις συζητήσεις με τους κοιόδης εισηγητές, όπου ο στόχος μας ήταν να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε εύστοχες και σύντομες προτάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να έχουν και απήχηση στο Συμβούλιο και να οδηγήσουν σε μια ταχεία έγκριση αυτού του θέματος. Παρ' όλα αυτά βέβαια πολλές φορές έχουμε καταθέσει υπερβολικό αριθμό τροπολογιών που θα πρέπει να τις επεξεργαστούμε και κάποια σημεία ίσως αυτή τη στιγμή έχουν ε, την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας ε, ώστε να γίνουν πιο ευανάγνωστα και πιο εύληπτα αλλά το έργο της κυρίας Ατζέα, της κυρίας εισηγήτριας ήταν ιδιαίτερα επιτυχίας για μας ως ΕΛΚ. Είναι πολύ σημαντικό, όπως ελέγχθη προηγουμένως, τα θέματα της, της πολιτικής αυτής ε, ε απασχόλησης να συνδεθούν με την πολιτική 20, Ευρώπης 2020. Ξέρουμε ότι οι συνδέσεις πολλές φορές δεν είναι παρούσες. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα ακολουθούν τους σημαντικότερους στρατηγικούς στόχους αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές και θα υπογραμμίσουν τη σημασία αυτών των στόχων από την άποψη αυτή. Πιστεύω ότι οι περισσότερες τροπολογίες μας κατευθύνονται προς την κατεύθυνση αυτή, στο σεβασμό της επικουρικότητας βέβαια, που πρέπει να είναι ένας σημαντικός παράγωνα και πολλές τροπολογίες ε, διαλαμβάνουν το θέμα των ε, αποδοχών, των συλλογικών συμβάσεων, των συνδικών εργασίας και είναι φυσικά και ο ρόλος των συλλογικών εστέρων, εταίρων μέσα στα κράτη-μέλη και θα πρέπει όλα αυτά να είναι ένα μέσο για την επίτευξη του σκοπού που έχουμε θέσει, αλλά θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτές οι προτάσεις θα μπορέσουν να τύχουν ε, ευήκοης ακρόασης, αλλά η προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται για την ε, αλλαγή των συνδικών δεν μπορούν να υποστηριχθούν από εμά. Κατά τα άλλα είναι μια θαυμάσια έκθεση, ήταν πολύ καλή συνεργασία των σχεδόν εισηγητών και πιστεύουμε θα είναι υποδομητικέ και υπεραιτέρω συζητήσει με του σχεδόν Ευχαριστώ πολύ. Μαρία Χάου Ροντρίγες. Χάου Ζουάου Ροντρίγες θα πρέπει να είναι εδώ αλλά δεν είναι εδώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μου ζήτησε η Μαρή Ζουάου να την εκπροσωπήσω. Θα ήθελα καταρχάς εκ μέρους της και θα ήθελα εκ μέρου τη ε, να συμφωνήσω με την αναγνώριση της ε, πολύ παραγωγικής ε, δουλειά της κυρίας Αγέα στην προσπάθεια εξέβρεσης συμβιβασμού με τρόπο που θα ενισχύσει τον ισχυρό χαρακτήρα του εγγράφου που θα μας δώσει έτσι μια ισχυρή θέση την οποία θα μπορούμε να παρουσιάσουμε. Ο σκιώδης εισηγητής ή ε, σκιώδης εισηγήτρια θεωρεί ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν καλό συμβιβασμό. Αυτό βασίζεται σε πολλές βελτιώσεις και επιτεύγματα τα ε, οποία ε, ήταν αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας με τους κοιόδης εισηγητές, την συμπερίληψη των στόχων ε, της στρατηγικής 2020, 20, ε, τα, τις απαιτήσεις που είχαν να κάνουν με τον ελάχιστο μισθό, καλύτερη διατύπωση σε σχέση με τη σύνδεση ελάχιστου μισθού και παραγωγικότητας, ε, σημαντικές μετατρομές, μετατροπές στη λειτουργία του, της αγοράς εργασίας, την ανάγκη ύπαρξη στρατηγικών επενδύσεων, ειδικότερα όσον αφορά τις δεξιότητες, ε, την ενίσχυση του ρόλου των βασικών δικτών και των ε, πινάκων των συγκριτικών, όπως επίσης και το θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ και της ε, διαρροής εγκεφάλων, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για την... και τα και την ε, καταπολέμηση της ένδυας. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι το τμήμα του συμβιβασμού είναι η στόχη της στρατηγικής 2020. Είναι αδύνατον ε, να τους, ε, να τους επιτύχουμε με τον τρόπο που αναφέρεται στη συγκεκριμένη έκθεση πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να αναφέρονται σιολογικές σκέψεις, πρέπει να είναι τμήμα των κατευθυντηρίων γραμμών που είναι κάτι ε, που ε, μας απασχολεί πολύ. Το πιστεύουμε ακράδαντα. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουν ε, σε μερικά σημεία, να αλλάξει μερικά σημεία και διατύπωση. Νομίζουμε ότι ο συμβιβασμός είναι πολύ καλός, ειδικότερα για τις μεταρρυθμίσεις συνταξιοδότησης και την σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης της νόμιμης με την δημογραφική αλλαγή. Ε, νομίζουμε ότι πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στην αύξηση της κοινωνικής επένδυσης, στην ενεργό γύρανση και επίσης αναζήτηση της αύξησης του ποσοστού απασχόλησης ως ενεργό αντιμετώπιση των προκλήσεων της, της γύρανσης του πληθυσμού. Σε γενικές γραμμές λοιπόν υποστηρίζουμε την εργασία της κυρίας Αγία και πιστεύουμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα καλό κείμενο. And now it's time for Mr. Once Ο κύριος Κρασνοντέμσκι. Αγγλικά θα τα πω ναι. αυτή τη φορά. να πω ότι εμείς είμαστε υπέρ των συμβιβασμών και θα ήθελα να πω ότι εκτός ε, από κάποια ζητήματα διατύπωσης ως ομάδα εμείς μπορούμε σε γενικές γραμμές να υποστηρίξουμε τους ε, συμβιβασμούς ε, που πρότεινε η κυρία Αγκαία και τις άλλες ομάδες. Υπάρχουν βέβαια κάποια προβληματάκια, γιατί και εμείς θα θέλαμε να τονίσουμε την άλλη πλευρά του προβλήματος, όχι μόνο την κοινωνική, αλλά και το πρόβλημα της ανάπτυξης και μιας πιο ενεργού πολιτικής ανάπτυξης. Να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα και εγώ να επενέσω την εισηγήτρια. Ήταν πάρα πολύ δραστήρια, πάρα πολλές συναντήσεις είχαμε μαζί της, μερικές φορές λίγο παράξενες, δεν είναι πάντοτε εύκολο να διαπραγματευτεί κανείς ε, την κάθε λέξη. Σας ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ ε, και είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε καλούς συμβιβασμούς ε, και πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα συμπορευτούν στους συμβιβασμούς αυτούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιος εκπροσωπεί τη Ρενάτε Βέμπερ από την ομάδα των φιλελευθέρων. Όχι, ο κύριος Ηλικιώτης τότε, εκ μέρους της Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την συνάδελφο την Λάουρα την Αιτζίαν ε, για την σκληρή δουλειά τη και την ειλικρινή συνεργασία. Ε, πράγματι έγιναν αρκετέ συναντήσει και υπήρχε ένα ανεπικοδομητικό πνεύμα. Εμεί ω GNGR συνεχίζουμε να είμαστε αισιόδοξοι για μια θετική κατάληξη για συμβαστικές τροπολογίες ε, και θεωρώ ότι μπορεί να, να καταλήξουμε σε μια πολύ καλή έκθεση αναφορικά με τις κατευθυντήρες γραμμές για την απασχόληση. Ε, θα ξαναπώ μερικά μόνο ζητήματα που θεωρούμε ότι ε, είναι αρνητικά σε αυτά που συζητούμε στην εκθεσή και βεβαίως καταθέτουμε πάντα τις απόψεις μας επικοδομητικά. Ε, και ιδιαίτερα στι συζητήσει για ε, τροπολογίε. <clears throat> Το πρώτο θέμα που μα απασχολεί έντονα και το έχω θέσει βέβαια στι είναι τα ζητήματα τη εκπαίδευση. Για μα είναι κέρια σημασία. Θεωρούμε πω η δημιουργικότητα, <clears throat> η καλλιέργεια κριτική σκέψη, η δημιουργία αντίληψη και και πρωτοβουλία στην εκπαίδευση δεν μπορεί να μεταφράζονται σε επιχειρηματικότητα από μικρή ηλικία. Δεν είναι συμβατά αυτά με την εκπαίδευση κατά ενόψη μα. Γι' αυτό εμεί θα προτιμούσαμε την αναθεώρηση των σημείων που, θεωρούν, ε, που προωθούν αυτή την προσέγγιση, την οποία θεωρούμε λαθασμένη. Επίσης, ε, η έννοια της αξιοπρεπούς διαβίωσης και της αξιοπρεπούς εργασίας, η οποία να σημειώσουμε καθορίζεται στην ατζέντα για αξιοπρεπή εργασία τη Διεθνή Οργάνωση για την Εργασία, των Decent World Agenda του ILO. Είναι πολύ σημαντικά και πραγματικά εκπλήττωνε, δεν κατανοώ πρέπει να πω, τη στάση ορισμένων, των εκπροσώπων ορισμένων πολιτικών ομάδων που θέλουν να διαγράψουν από την έκθεση αυτέ τι εκφράσει. Δηλαδή την έννοια της αξιοπρεπής διαβίωσης και της αξιοπρεπούς εργασίας ε, που θεωρούμε είναι σημαντικές όταν μιλούμε ε, για, την, ε, για τις κατευθύνσεις, καθυντήρες γραμμές για την απασχόληση. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την εσωμάτωση αυτής της έννοιας στο κείμενο. Τέλος, αναφορικά με τη μεταφορά της φερολόγησης από την εργασία. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε το κείμενο, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να δούμε ελάφρυνση της φορολόγηση των εταιριών αναφορικά με το εργατικό κόστος αν αυτήν την ελάφρυνση θα την επιμοστούν οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι καταναλωτές, τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα μέσω των έμμεσων φόρων. Για μα είναι σημαντικό η φορολογία για την εργασία να διανέμεται δίκαια και με αναλογία μεταξύ των μεγάλων και των μικρών επιχειρήσεων και των κερδών του, χωρίς να απειλείται με τέτοια μέτρα η κοινωνική προστασία των εργαζομένων ή να χρειάζεται να πληρώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τη μερίδα δηλώνοντος για την κοινωνική και την εργασιακή τους ε, ασφάλιση. Και πάλι ολοκληρώνω λέγοντας ότι ε, θεωρούμε ότι μπορεί να καταλήξουμε ε, σε ένα θετικό κείμενο και να συγχαρώ ακόμα μια φορά την συνάδελφο τη Λάουρα για την δουλειά της. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you, Madam Stanoka. Η κυρία Στανοκα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς αρχικά ήμασταν ανικανοποιητοί με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, απόφαση του Συμβουλίου σε σχέση με τις κατευθυντήρες γραμμές και είναι ακόμα λιγότερο φιλόδοξο το κείμενο αυτό από ό,τι περιμέναμε. Γι' αυτό ήταν ένα τιτάνιο έργο για την εισηγητριά μας να μπορέσει να καταλήξει μια καλή εκθέση για τις γραμμές. Το τέτοιο όμως αυτό και πρέπει να εκτιμήσω, να εξάρω ιδιαίτερα το έργο της κυρίας Αγίας. Και η ομάδα μας έχει καταθέσει μια σειρά από τροπολογίες και ο μεγάλος αριθμός των τροπολογιών είναι απάβγασμα του, των προτάσεων της Κομισιόν και της ασάφειάς τους που δεν έχουν παρά μόνο γενικό χαρακτήρα δηλώσεων πρέπει όμως να τις συγκεκριμενοποιήσουμε και αυτός είναι ο στόχος των συνεδριάσεων των σκιωδών εισηγητών και των τροπολογιών συμβιβασμού ώστε να πάμε προς την σωστή κατεύθυνση παραδείγματος παραδείγματος χάρη δεν επαρκεί η απλημνία της στρατηγικής Ευρώπης 2020 και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει να ξέρουμε πιο συγκεκριμένα τι θέλουμε να κάνουμε, τι θέλουμε να επιτύχουμε. Παραδείγματος στις αιτιολογικές σκέψεις θέλουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τις προσπάθειες που έχουν να κάνουν με τη μείωση των ανισοτήτων εισοδημάτων μεταξύ των πολιτών. Αυτός πρέπει να είναι τους κέριους στόχους μας και να αντιμετωπίσουμε την ένδυα και, και τον κοινωνικό αποκλεισμό Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν αυτές τις στρατηγικές όπως και τη στρατηγική εκπαίδευση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, είναι στόχοι αλληλένδετοι και αλληλοενισχυόμενοι στόχοι. Οπότε επίσης εδώ πέρα αναφερόμαστε σε καταληκτικές προθεσμίες και πολιτικές των κρατών μελών. Το πιο σημαντικό εδώ είναι να δούμε τι θα κάνει και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το πλαίσιο και θα θέλαμε περαιτέρω να υπογραμμίσουμε εδώ ότι τα κράτη-μέλη όταν δέχονται κάποιες οικονομικές πολιτικές αυτό πρέπει να το κάνουν με κοινή συνένεση και θα πρέπει να γίνεται με συντονισμό και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. και απομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνδυάζει αυτές τις διατάξεις με προτάσεις για την επίτευξη των στόχων της συνθήκης, κάτι το οποίο συμπεριλαμβάνει και καλύτερε συνθήκε εργασία και ολοκληρωμένη αγορά εργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητο ω εκ τούτου οι πολιτικές αυτές τη Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην τίθενται εν αμφιβόλο και γι' αυτό έχουμε καταθέσει σχετικές τροπολογίες προς την κατεύθυνση τροπολογιών συμβιβασμού. Πολλή δουλειά έχουμε να κάνουμε ακόμα και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε ένα πολύ καλό κείμενο. Ελπίζω θα ευδοκιμήσουν όλες αυτές τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση εκθέσεως μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ανεφέρθη η Κομισιόν. Υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν ο οποίος θα ήθελε να προσθέσει κάτι σχετικά. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε σημειώσει τις τροπολογίες, έχουμε πάρα πολύ, με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθήσει το σχέδιο γνωμοδότησης και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θέλω απλώ να πω ότι η έγκριση στην Επιτροπή μας ε, θα γίνει στις 16 Ιουνίου. Πάμε στο σημείο 19 της σημερινής διάταξης. Πράσινη απασχόληση, αξιοποίηση των δυνατοτήτων ε, της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας είναι η πρώτη ανταλλαγή ε, απόψεων για τις τροπολογίες 208 τον αριθμό συνολικά για την γνωμοδότηση της κυρίας Λάμπερτ και θα ήθελα να της δώσω το λόγο. Έχετε το λόγο κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Αναφερθήκατε στον αριθμό των τροπολογιών ε, για την ε, έκθεση αυτή. Ε, ε, ελπίζω ο λόγος να είναι διαφορετικός. Οι περισσότερες τροπολογίες είναι θετικές και οι γενικές γραμμές προσπαθούν να προσθέσουν σε αυτό που είχαμε συμπεριλάβει στην αρχική έκθεση και νομίζω ότι οι περισσότερες είναι πολύ επικοδομητικές και μπορούμε πολύ καλά να τις ενσωματώσουμε. Το ιστορικό είναι το εξής η ανακοίνωση της Επιτροπής που αναφέρθηκε σήμερα το πρωί από τον Επίτροπο Ντομπρόφσκης. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε σαφή στρατηγική, σαφή μηνύματα πολιτική, συνοχή για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας, όχι μόνο σε όλους τους τομείς, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούμε τις αλλαγές εντός ορισμένων τομέων, που μπορεί να είναι πάρα πολύ ε, ρηπογόνη, είναι υπεύθυνη για πολλές ε, εκπομπές αερίων και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την αλλαγή. Πρέπει να πω ότι προσπαθώ να βρω έναν ευγενικό τρόπο να το πω, ήμουν κάπως απογοητευμένη με την ανταπόκριση της, ε, του Επιτρόπου σήμερα το πρωί ε, στην απάντησή του όταν τον ρωτήσαμε για το πώς εντάσσεται αυτό στη στρατηγική απασχόληση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς θεωρούν ότι μπορεί να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και αν αποτελεί σαφή φιλοδοξία ε, ή απλώς ε, μια αναγνώριση της κατάστασης. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές οι τροπολογίες είναι πάρα πολύ επικοδομητικές, θετικές. Είχαμε γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και από την Επιτροπή Γυναικών ε, και οι δύο επιτροπές ε, πάρα πολύ σημαντικά σημεία θέτουν. Ε, υπάρχουν βέβαια και κάποιες αλληλοεπικαλύψεις, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εντάξουμε αυτές τις βασικές ιδέες που προέρχονται από τις γνωμοδοτούσες επιτροπές αυτή τη στιγμή εργάζομαι επί του συμβιβασμού. Ε, χτες είχαμε μια εισαγωγική συνάντηση για να γίνει μια πρώτη εξέταση. Θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις, το έχω υποσχεθεί. Σήμερα το πρωί για την κυκλική οικονομία και με την ψηφοφορία μας δείξαμε ότι έχουμε μια συγκεκριμένη ε, σχέση με το θέμα, γιατί το θέμα της κυκλικής οικονομίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχουν ε, σχέσεις και ε, σύνδεσμοι με αυτό που συζητούμε τώρα. Δύο-τρεις ε, τομείς, τους οποίους θεωρούμε ότι έχουμε διαφορετικές οπτικές γωνίες. Παράγραφος 14 είναι μία από αυτούς τους τομείς. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για το ρόλο των κινήτρων και νομίζω το θέμα είναι η δεσμευτική στόχοι. Μπορεί να βρούμε μια συμβιβαστική λύση η οποία δεν αναφέρει συγκεκριμένα τους δεσμευτικούς στόχους αλλά μπορούμε να ψηφίσουμε κάποιους τροπολογίες όπως για παράδειγμα την 131 της ΓΚΟΕ οι οποίες ε, έχουν συγκεκριμένες αναφορές ε, για συγκεκριμένους στόχους και πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις βασικές αυτές ιδέες και μετά να δούμε πώς ε, μπορούμε να ε, κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα δεύτερο τομέα ένα δεύτερο τομέα είναι η παράγραφος 16 για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη νέα οδηγία περί προμηθειών, ειδικότερα ε, στην κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση και πόσο θέλουμε να το πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αναμένω σχόλια από τους συναδέλφους κατά πόσο η 143 τροπολογία του κυρίου Μαν η οποία είναι κάπως πιο διερευνητική προς αυτή την κατεύθυνση, κατεύθυνση να ε, εξετάσουμε δηλαδή κατά πόσο είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Η άποψή μου είναι ότι ναι, όντως είναι ένας τρόπος. Ελπίζω να συμφωνήσουμε και ίσως και κάποια σημεία τα οποία η Επιτροπή των Περιφερειών μου είπε στην τροπολογία τη δική μου 155 αποσαφήνιση ορισμένων ε, παραγόντων αυτής της οδηγίας για τις προμήθειες. Ελπίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Παράγραφος 18 και η αιτιολογική σκέψη F πάλι αποτελεί ένα τομέα διαφιλονικού, ενώ ειδικότερα όταν βλέπουμε το όταν βλέπουμε ε, για το όταν βλέπουμε την ε, σχέση της κυκλικής οικονομίας με την αγορά εργασίας, είναι κάτι το είδαμε και σήμερα το πρωί, το ψηφίσαμε, η, η μεταφορά της φορολογίας ε, περισσότερο από την εργασία και πιο πολύ προς τη μεριά του περιβάλλοντος. Ίσως αυτό ε, να ήταν μία λύση. Νομίζω ότι οι σοσιαλιστές και οι γκου έχουν προτείνει τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Η άποψή μου είναι ότι όντως αυτό αποτελεί ένα τμήμα των κινήτρων ε, για τις επενδύσεις του συγκεκριμένο τομέα και βέβαια δημιουργία θέσεων απασχόλησης και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συμφωνήσουμε για το πώς θα το πούμε αυτό. Άλλους τομείς στους οποίους νομίζω συμφωνούμε περισσότερο ε, είναι θέμα διατύπωση μόνο. Το θέμα της διάστασης ε, του φύλου, αυτό προέρχεται από τη γνωμοδότηση Επιτροπής των Γυναικών, πώ θα μπορέσουμε να το λάβουμε αυτό υπόψη, η 117 τροπολογία του κυρίου Κέλλερ επίση, να είναι σαφέ ότι αν υπάρξουν νέε θέσει απασχόληση ή αλλαγές στο χώρο εργασίας, θέλουμε να απομακρυνθούμε από αυτήν την τομεακή διάσταση γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ε, για πολύ μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των φύλων και κάλυψη του χάσματος των αμοιβών ε, μεταξύ των δύο φύλων ε, στο πλαίσιο εξωπρεπούς εργασίας πάντοτε. Πάρα πολλές χρήσιμες τροπολογίες υπήρξαν επίσης επί ειδικών προτάσεων για τις δεξιότητες και την ανάπτυξη αυτών που μπορούμε νομίζω να τις συγκεράσουμε με την 197 τροπολογία και νομίζω και η 98 και η 100 τροπολογία πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι είναι ε, πάρα πολύ ισχυρές και αφορούν τις δεξιότητες. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε. Μας δίνει μία αίσθηση της κατεύθυνσής μας έχουμε πολλές δυνατότητες, πρέπει να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη μετάφαση, να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ότι υπάρχουν τα σωστά κίνητρα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρομεσαίες, ε, ε, το ανέφεραν αυτό και κάποιες τροπολογίες, να μπορέσουν να μας ε, δώσουν όλες τις δυνατότητες που, που μπορούμε να έχουμε στο πλαίσιο της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Και δεν μιλάμε μόνο για τις πιο συμβατικές θέσεις εργασίας, προσπαθούμε να βρούμε πώς μπορούμε να εξελιχθούμε από αυτό και από κοινωνικής και από περιβαλλοντικής απόψεως. Με μεγάλη χαρά θα ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτή την πολύ επικοδομητική ατμόσφαιρα που υπήρχε ως τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κλούνες και η του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστώ και την κυρία Λάμπερτ για τα σχόλιά της. Είχαμε μια πρώτη συνάντηση σκιωδών χθες. Και πολλά από τα σχόλιά μας ήταν περισσότερο προστίκες παρατροποποίησης για να συμπληρώσουμε την αρχική ανακοίνωση της Κομισιόν. Εγώ θα είχα κάποιες προτάσεις να κάνω και τροπολογίες σε σχέση με το χάσμα δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να αναφερθεί. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την ανάπτυξη προσόντων και δεξιοτήτων και συστήματα όπως η Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστώσουμε τα κενά ε, δεξιοτήτων και οι πράσινες δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε και μεγαλύτερη διακινητικότητα μέσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε πού υπάρχουν κενέ θέσει και πού θα αναπτυχθούν και πού λοιπόν μπορούμε με το σύστημα αυτό να έχουμε ένα ρόλο για να εξασφαλίσουμε καλύτερη κάλυψη των θέσεων τη πράσινη οικονομία. Όπω είπε η κυρία Λάμπερτ, υπάρχει τεράστιο δυναμικό στι μικρομεσαίε επιχειρήσει για την πράσινη οικονομία για να δημιουργήσουν θέσει εργασία στον τομέα τη ε, απομόνωση των κτηρίων, τις πράσινες τεχνολογίες, την λεγόμενη κυκλική οικονομία, την ανακύκλωση. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να επιτευχθούν λοιπόν χάρη στην πράσινη οικονομία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό τμήμα της εκθέσεως την οποία θα συντάξουμε σε σχέση με άλλους τομείς. Υπάρχουν κάποια σημεία ίσως τριβής τα οποία μπορούν να προκύψουν σε ό,τι αφορά την ε, μετακίνηση της φορολογίας προς την ε, απασχόληση. Εμείς θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να προκύψει για χαμηλής δεξιότητος ε, θέσεις απασχόλησης. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε για το θέμα μετακίνησης, μετακύληση της φορολογίας από την εργασία στο περιβάλλον και επίσης για τους δεσμευτικούς ε, στόχους πρέπει να έχουμε νομοθεσία, αλλά η νομοθεσία αυτή δεν θα πρέπει να είναι μοναχα νομοθεσία για την νομοθεσία, θα πρέπει να είναι νομοθεσία για την καλύτερη νομοθεσία. Αυτά τα σημεία λοιπόν μπορούμε ίσως να τα διευκρινίσουμε καλύτερα μαζί με την εισηγήτρια. Η κυρία Λάμπερτ έχει ένα δύσκολο έργο για να μπορέσει να καταλήξει σε συμβαστικέ λύσει, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρει και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί τη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Γιάνν από λιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε μια έκθεση η οποία ασχολείται με τις λεγόμενες πράσινες θέσεις εργασίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην έχουμε δημιουργία οποιασδήποτε θέση εργασίας, αλλά μια θέση εργασίας η οποία έχει ποιότητα αυτό, πρέπει να το δούμε από διάφορες πτυχές πρώτα απ' όλα. Τονίζουμε την ανάγκη να υπάρξει κοινωνικός διάλογος. Ο κοινωνικός διάλογος στον τομέα αυτό φαίνεται πολλές φορές να είναι απόν. Και είναι σε ορισμένα κράτη ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, διότι τα συνδικάτα είναι από τους μεγαλύτερους αντιπάλους της δημιουργίας πρασίνων θέσεων απασχολήσεως. Γιατί, το λέω αυτό γιατί έχω εργαστεί εδώ και πολύ καιρό με τα εργατικά συνδικάτα. Είναι πάντα ιδιαίτερα επιφυλακτικές εργατικές ενώσεις σε ό,τι αφορά τις πράσινες θέσει εργασίας, όχι ότι δεν είναι οικολόγοι. Αλλά πολλές φορές αυτά οδηγούν στο να εξαφανίζονται καλοπληρωμένες θέσεις συμβατικής εργασίας στη βιομηχανία και οδηγεί στην ανάδυση νέων θέσεων εργασίας που είναι λιγότερο ε, ασφαλής από κοινωνική άποψη και λιγότερο καλοπληρωμένες. Επομένως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πράσινες θέσεις εργασίας είναι θετικού χαρακτήρα. Δεύτερον, το στοιχείο των πρασίνων θέσεων εργασίας είναι πολλές φορές θηλυκοποιημένου χαρακτήρα. Αφορούν τις γυναίκες. Καλό είναι οι γυναίκες να έχουν ίσα δικαιώματα εργασίας και να είναι εξισωμένες με τους άνδρες στον τομέα εργασίας. Αλλά όταν θέλουμε να έχουμε ε, θέσεις εργασίας με τις πράσινες τεχνολογίες πρέπει να προσέχουμε γιατί οι εργασίε αυτέ απευθύνονται κυρίω σε γυναίκε και είναι χειρότερα πληρωμένε. Και ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά τις χαμηλές αποδοχές, εκεί μονάχα υπάρχει ισότητα ανδρών και γυναικών. Γι' αυτό και πάλι τονίζω ότι πρέπει αυτές τις εργασίες να είναι αξιοπρεπείς και υψηλής ποιότητας. Και τρίτον, σε ό,τι αφορά την μετάβαση από την φορολογία της εργασίας στην ε, φορολογία των αρνητικών εξωτερικοτήτων του περιβάλλοντος, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εδώ μπορούμε να καταλήξουμε σε απαγορευτικού ύψους φόρους. Για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί θα πρέπει να αποφύγουμε να μειωθεί και η δυνατότητα εξασφάλιση των θέσεων εργασίας. Να μην δημιουργηθούν μονάχα επισφαλείς θέσεις εργασίας, αυτό θα είναι μια πραγματική απειλή κατά της πράσινης οικονομίας γιατί θα σημαίνει ότι η πράσινη οικονομία οδηγεί κατευθείαν στην ένδια. Αυτό δεν θα βοηθήσει ούτε τις γυναίκες, θα εξοργήσει τα συνδικάτα. Εν πάση περιπτώσει εγώ θα υποστηρίξω τις ε, συμβαστικές τοπολογίες που έχει προτείνει η κυρία Λάμπερτ και εγώ υποστηρίζω ότι θα πρέπει να εισαχθούν και δεσμευτικοί στόχοι πρόκειται για ένα νευραλγικό τομέα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα σώσουμε τη γη, αλλά αυτό γίνεται με εθελοντικά μονάχα μέτρα. Οι στόχοι μας θα πρέπει λοιπόν να υποστηριχθούν με δεσμευτικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλερ. Υπάρχει κάποιος από την ομάδα των φιλελευθέρων. Όχι. Από τη συντηρητική ομάδα. Όχι. Η Λίν Μπόιλεν από ο κύριος Ηλικιώτης εκπροσωπεί την κύριε Μπόιλεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, αναπληρώ, αντικαθιστώ την σκιώδη εισηγήτρια από την QNGL, την Λίν Μπόιλεν. και πρέπει να πούμε ότι εμείς καλωσορίζουμε τις συμβαστικές τροπολογίες και ευχαριστούμε την εισηγήτρια την κυρία Λάμπερτς για την καλή και επικοδομητική δουλειά. Είμαστε τη άποψη πω είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τι αναφορέ στην ατζέντα για την αξιοπρεπή απασχόληση στην έκθεση για την πράσινη απασχόληση. Ω Επιτροπή Απασχόληση του Κοινοβουλίου πρέπει να τονίσουμε πω αυτέ οι πράσινε θέσει απασχόληση πρέπει να είναι αξιοπρεπεί, διασφαλισμένε και καλοπληρωμένε. Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια άλλων ομάδων να διαγράψουν τι αναφορέ σε αξιοπρεπεί και ασφαλεί θέσει εργασία. Ε, η ομάδα μα καλωσορίζει τη συμβαστική τροπολογία αριθμό 4 αναφορικά με τον ρόλο των εργαζομένων στη μετάβαση για μια πράσινη οικονομία. Είμαστε τη άποψη πω οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα του έχουν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση η οποία πρέπει να λάβει χώρα κάτω από τα κάτω, δηλαδή το επίπεδο του χώρου εργασίας προς τα πάνω, δηλαδή το εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή μα πρέπει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην έκθεση πω θέλουμε να δούμε του εργαζόμενου και τα συνδικάτα του βαθιά αναμειγμένου σε όλα τα επίπεδα αυτή τη διαδικασία. Αναφορικά με το θέμα των περιβαλλοντικών φορολογιών, έχουμε ανησυχίε σε σημεία τη πρόταση τη Επιτροπή. Εν τούτης, ε, δεν είμαστε αντίθετοι με την αρχή πω οι μεγάλοι ρηπαίνοντε πρέπει να πληρώνουν για τι ενέργειέ του. Η ανησυχία μας εστιάζεται στο γεγονός ότι κάποιοι φόροι που θα εισαχθούν στα κράτη-μέλη και οι οποίοι ονομάζονται περιβαλλοντικοί δεν στοχεύουν τελικά τους μεγάλους ρηπαίνοντες αλλά επιβάλλουν αναδρομικούς φόρους για τους καταναλωτές και πλήττουν σκληρότερα τα πιο φτωχά στρώματα της κοινωνίας εφόσον είναι ισοπεδωτικοί φόροι. Είμαστε της άποψης πως αυτή η διάκριση πρέπει να υπογραμμιστεί στην εκθέση. Τέλο, αναφορικά με το ζήτημα των δημόσιων συμβάσεων, η ομάδα μα στηρίζει στεναρά την πρόταση που έγινε στην έκθεση τη Επιτροπή ότι οι δημόσιε συμβάσει θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενεργητικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο το οποίο μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά και να καθοδηγήσει κυβερνήσεις κρατών μελών στο να συνεισφέρουν στην κοινωνική δικαιοσύνη και στο περιβάλλον κατά τις διαδικασίες των συμβάσεων. Ολοκληρώνοντα και πάλι να συγχαρώ την εισηγήτρια την κυρία Λάμπερ για τη σκληρή δουλειά που κάνει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank you. Laura Agia. Ευχαριστώ. Η Λάβρα Αγία από το EFTD. Ε, Σα ευχαριστώ και πάλι κυρία Πρόεδρε και θέλω απλά να πω ότι Συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που προτάθηκαν, δηλαδή συμβιβασμοί που διατυπώθηκαν από τη συνάδελφο Τζιν Λάμπερτ. Πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχει αναφέρει με τη μορφή των συμβιβασμών και εμεί θα θεωρούμε όλα αυτά πολύ σημαντικά. Και επίσης ε, θεωρούμε ότι είναι και πολύ σωστό ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δική μας η πρόταση, η δική μας η τροπολογία, εκεί όπου ζητάμε να υπάρχουν κέντρα έρευνας που θα ε, παρουσιάζουν νέα προγράμματα, νέες τεχνολογίες, ε, νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ε, άρα δηλαδή πράσινη τεχνολογία. Και αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να υιοθετηθεί από τις πράσινες επιχειρήσεις γιατί η απασχόληση εκτός από θέματα ποιότητας η απασχόληση έχει να κάνει και με περιβαλλοντικά θέματα όπου λοιπόν δεν υπάρχει η αηφορία και όπου δεν λαμβάνεται υπόψη το στοιχείο του περιβάλλοντος νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα είμαστε αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουμε έναν πλανήτη ο οποίος ε, θα μας ε, ζητήσει τον τελικό λογαριασμό. Σε γενικές λοιπόν γραμμές ε, συμφωνούμε με τη συνάδελφο στην πρώτη συνάντηση των ε, σκιωδών ε, συντονιστών, προχθές δηλαδή έγινε αυτό, είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες ε, δυσκολίες όσον αφορά τη μετακύληση της φορολόγησης. Νομίζω ότι παρόλα αυτά είναι σημαντικό να χαράξουμε μια αποτελεσματική πολιτική και θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπα και προηγουμένως. Δηλαδή πράγματι να υπάρχει μια πράσινη οικονομία η οποία μέχρι κάποιου βαθμού ε, θα επιτρέπει να ε, αποκαθίστανται οι ε, ζημιές. Οι ζημιές που προκαλούνται από υπερβολική παραγωγή, υπερβολική δόμηση, πολλά, πολλές φορές αυτά προκαλούν ζημιές και το θέμα είναι ότι να μην ασχολούμεθα μόνο με την αποκατάσταση, δηλαδή εξέβρεση εργασίες εργασία σε ανθρώπους, αλλά αποκατάσταση και ενταφών και εκτάσεων. Κατόπιν τούτου, αυτά θα πρέπει να τα έχουμε κατά νου, κυρίως τώρα, κατά την περίοδο της κρίσης. Η πράσινη απασχόληση ε, νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ίσως είναι ο μόνος ε, οικονομικός τομέας ο οποίος ε, έχει ακόμα τη δυνατότητα να προσφέρει εγγυήσεις για αυτές τις θέσεις που ήδη υπάρχουν. Επίσης, πολύ σωστό και αυτό που ελέγχθη σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων, δηλαδή να υπάρχει ίση ίσες, να υπάρχουν ίσες απολαμβές ε, για, τον, για την ίδια εργασία. Αυτό απαιτεί βέβαια μία σειρά μέτρων που όμως κρίνονται απολύτως απαραίτητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Την εισηγήτρια και τις σκιές που την περιστοιχίζουν η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας είναι στις 16 Ιουνίου και στο μέλια το Σεπτέμβριο. 2015. Θέμα υπαριθμών 20 τελευταίο, όχι ίστατο όμως, μονοπρόσωπες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένες ευθύνες. 245 και μόνο τροπολογίες έχουν κατατεθεί για την νομοθετική πρόταση της οδηγίας που θεσπίζει μονό προσωπικές ε, περιορισμένες ευθύνες εταιρείε. Είναι μια έκθεση της Επιτροπής Γιούρι και εμείς βάσει του 54 ζητήσαμε να συμμετάσχουμε μαζί με την Επιτροπή Γιούρι. Απέτυχε όμως αυτό γιατί δεν το δέχτηκε η συνέλευση των Προέδρων. Δίνω το λόγο στην κυρία Στάινρουκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μπορώ να είμαι σχετικά σύντομη. Την προηγούμενη εβδομάδα συναντηθήκαμε με τους σκιώδεις εισηγητές και συζητήσαμε για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις τροπολογίες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Έχουμε συμφωνήσει και σε μεγάλο βαθμό έχουμε καταλήξει σε μια συνένεση να ε, απορρίψουμε κάποιες ε, συμβαστικές τροπολογίες. Είπαμε ότι δεν είναι απαραίτητο να έχουμε συμβαστικές τροπολογίες τη στιγμή που τα πράγματα είναι σαφή. Περιμένουμε λοιπόν από την Κομισιόν να καταλήξει σε νέες προτάσεις, τις οποία, τις οποίες προτάσεις θα λάβει υπόψη και τις αιτήσει των πολιτικών ομάδων. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο εμείς θέλουμε να δώσουμε προς το παρόν από την δική μας πλευρά. Ευχαριστώ. Από το ΕΛΚ. Ναι. Εκπροσωπώ τον συνάδελφο, τον κύριο Κάζα. Το ΕΛΚ πάντοτε συμφωνούσε με την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα μέτρα διευκόλυνσης του εμπορίου τους ε, και αυτή η νομοθεσία σκοπό έχει να καταστήσει ευκολότερα τα πράγματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμφωνούμε όταν βλέπουμε τώρα τον αντίκτυπο υπάρχουν πολλά ζητήματα που μας απασχολούν, όπως για παράδειγμα ότι θα μπορούσαμε να δημιουργούμε ε, εταιρείε χαρματοκιβώτια ε, και υπάρχουν και τα προβλήματα προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι κάθε εργαζόμενος προστατεύεται. Αυτή η νομοθεσία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επιβλαβείς συνέπειες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι, το, η, ότι η συγκεκριμένη έκθεση θα έχει ως αποτέλεσμα την ε, προστασία των ε, εργαζομένων και θα θέλαμε να προτείνουμε την απόρριψη της συγκεκριμένης πρότασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κροσεντέμσκι. Θα μιλήσω γερμανικά έτσι από αθλητικό πνεύμα. Ήθελα να πω ότι καταρχήν η ιδέα είναι θετική. Και την έχουμε υποστηρίξει την ιδέα αυτή να υπάρχει η δυνατότητα πιο εύκολα να μπορεί κανείς να συγκροτεί εταιρείε οι οποίες μπορούν να δουλεύουν διαμεθοριακά και αυτό ευνοεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δυστυχώς, δυστυχώς υπάρχουν πολλές ανησυχίες που έχουν παραμείνει και δεν έχουν διασαφινιστεί από την πλευρά της Κομισιόν. Πολλοί μου έθεσαν ερωτήματα, παραδείγματος χάρη, μεταξύ της, ε, η διάκριση μεταξύ της έδρας της επιχείρησης και της έδρας καταχώρησης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα και γι' αυτό την απορρίπτουν οι περισσότεροι συνομιλητές μου. Και γι' αυτό κρατάμε μια πολύ επιφυλακτική στάση. Ίσως θα μπορούσε να υπάρξει από την πλευρά της Κομισιόν μια καλύτερη πρόθεση. Ευχαριστώ και μερσή λέει πρόεδρος. Από την ομάδα της Άλντε υπάρχει κάτι που θέλει να λάβει το λόγο. Όχι. Από την Γκούε ούτε. Μετά θα πάμε στους πράσινους. Όχι. Ούτε και εσείς κύριε Λάμπερτ. Η κυρία Τζέα. Ξέχασα κάποιον, την κυρία Τζέα. Α, τη Λαύρα. Έχετε το λόγο. brevissima. Ma in realtà io parlo Κοιτάξτε, εγώ ομιλώ εξ ονόματος της αδέλφου Μπεγκίν, που ε, και αυτή έχει τις ίδιες ακριβώς ανησυχίες. Είχε προετοιμάσει μια παρέμβαση. Ε, τέτοια πράγματα λέμε και δεν θέλω να καθυστερήσω περισσότερο τη συζήτηση. Όπως ε, είπε και η συνάδελφος ε, εκ μέρους του κυρίου Κάζα, το θέμα είναι ότι με τον τρόπο αυτό ε, ευνοούνται παράνομοι και μη διαφανείς μηχανισμοί. Άρα συμφωνούμε απόλυτα με αυτό που προτείνει η κυρία να απορριφθεί αυτή η πρόταση. Thank you. Are there any... Merci, λέει η πρόεδρος. Υπάρχουν κάποιος από την Κομισιόν που θέλει να σχολιάσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Νομίζω ότι απλώς πρέπει να καταγράψουμε την αρνητική αυτή θέση της Επιτροπής σας. Ακούσαμε και φήμε, φήμες από τις συνεδρίες του Συμβουλίου για το θέμα αυτό αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Οκ. Okay. Τούτου λεχθέντος. Η έγκριση στην Επιτροπή Απασχόλησης θα είναι στις 23 Ιουνίου, στην Επιτροπή Γιούρι στις 15 Σεπτεμβρίου, τούτων λεχθέντων έχουμε φτάσει το τέλος και την πλήρη εξάντληση στη συνεδρίασή μας. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 15 και 16 Ιουνίου στις ίδιες αυτές Βρυξέλλες και σας ευχαριστώ τα μάλα για τις τόσο ενδιαφέρουσες συζητήσεις και εκθέσεις και καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.